συνεδρίασης σας διανεμήθηκαν. Δεν ξέρω κατά πόσο να έχετε αντιρρήσεις επ' αυτών. Από ό,τι βλέπω όχι. Ε, κατόπιν τούτου ε, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη θα έχουμε τις δηλώσεις ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά ε, να μπορούμε να καλωσορίσουμε εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας, ε, τον κύριο Σβάτσενμπερκ, ο οποίος σήμερα το βράδυ θα πάει στη Νότια Αφρική και οι ε, παλαιότερες ε, προεδρίες έκαναν το εξής. Δεν ερχόντουσαν οι ίδιοι Υπουργοί Εξωτερικών, έστελαν τους αντικαταστάτες τους. Γι' αυτό ε, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Σφάτσενμπερκ για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα εδώ. Έχουμε και την κυρία Μπενίτα Φερέρο Βάλτνα, την αρμόδια επίτροπο η οποία επίσης γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Μέσης Ανατολής και η ίδια έχει ήδη πάει επί τόπου, όπως και ο κύριος Σφάτσεμπερκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγοι είμαστε εδώ, λίγοι αλλά καλοί. Ε, ενδιαφερόμεθα όλοι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό ε, και παρακαλώ τον κύριο Σβάτσενμπερκ να ε, λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο αυτή την ώρα των ε, συζητήσεων ως προς τη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κύριε Πρόεδρε, από την έναρξη της ε, προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές στο Ισραήλ βλέπουμε ότι επιδεινούνται η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Οι ανθρωπιστικές συνέπειες αυτού του εγχειρήματος είναι δραματικές για τον πληθυσμό της Γάζας. Από την ε, αρχή των επιχειρήσεων 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί ενώ το 30% είναι άμαχος πληθυσμός, γυναίκες και παιδιά. Μας ε, λυπεί ιδιαίτερα αυτή η απώλεια και ξέρετε ότι έχουν γίνει επαναλημμένες δηλώσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για, τις ε, συνεχόμενες, για τη συνεχόμενη σύραξη που έχει οδηγήσει σε σκοτωμό του άμαχου πληθυσμού και έχουμε αποστείλει τα συλληπιτήρια στις οικογένειες και επίσης Δυστυχώς σκοτώθηκαν πολλά παιδιά στο σχολείο, σε ένα σχολείο των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν τραυματιστεί 4.200 Παλαιστίνοι, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. και 28.000 έχουν μετατοπιστεί από την αρχή των εχθροπραξιών. Ε, και πολλοί προσπαθούν να μεταφερθούν στα καταφύγια. Υπάρχουν μεγάλες ανθρωπιστικές ανάγκες και οι υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να ανταποκριθούν μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και δίδοντας καταφύγιο στον ε, άμαχο πληθυσμό. Το υδροδοτικό σύστημα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και γι' αυτό ακριβώς ο πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι ύψης της σημασίας. Επίσης υπάρχουν ε, ελλείψεις τροφίμων σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού. Από τις 4 Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους πολλές μη κυβερνητικέ δεν μπόρεσαν να μεταβούν στη Γάζα για να αντιμετωπίσουν το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Επίσης, πολλοί Ισραηλινοί έχουν ε, μεταβεί μέσα στα πλαίσια των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές και μπόρεσαν να εισχωρήσουν στο έδαφος μόνο 300 φορτηγά προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τα τραγικά γεγονότα από την αρχή. Τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συνήλθαν στο Παρίσι για να εξετάσουν την έκτακτη κατάσταση και έκριναν ότι θα πρέπει να δοθεί άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και να αποκατασταθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να λήξει η βία. Η Προεδρία λοιπόν ανέλαβε μία διπλωματική αποστολή στη Μέση Ανατολή. Επισκεφθήκαμε την ε, περιοχή από τις 4 έως 6 Ιανουαρίου για να συναντηθούμε στην Αίγυπτο και στην Ιορδονία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Επίσης, ο επισκεφθήκαμε την Συρία, το Λίβανο και την Τουρκία. Βλέπουμε την απαρχή μιας λύσης και θεωρούμε ότι καταρχήν η Χαμάς θα πρέπει να σταματήσει την ρήψη πυράβλων στο Ισραηλινό έδαφος και επίσης να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και οι Ισραηλινοί έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης ε, χρειάζονται Χρειάζεται ιατρική υπερηθαλψή. Στις 19 Δεκεμβρίου έληξε η ανακοχή, αλλά δεν ήταν η ιδεώδης. Δυστυχώς ερήφθησαν πολύ πύραυλοι στο Ισραηλινό έδαφος και κατά τη διάρκεια και της, της εκεχηρίας από την Χαμάς. Επίσης η Γάζα είχε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση οικονομικού αποκλεισμού. Για να φτάσουμε σε μια βιώσιμη εκεχηρία θα πρέπει να φτάσουμε σε έναν λογικό συμβιβασμό και να σταματήσουν οι ρήψεις πυράβλων. Μια βιώσιμη λύση θα πρέπει να είναι διασυνοριακή και επίσης θα πρέπει να ανοίξουν όλες οι διελεύσεις των συνόρων για να μπορέσει η Γάζα να ανατροφοδοτηθεί. Τροφοδοτηθεί, με συγχωρείτε. Θα πρέπει να προωθηθεί λοιπόν η εκεχηρία και υπ' αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να αποστείλει παρατηρητές στη Ράφα εκ νέου και να παρατείνει την εντολή της αποστολής στα σύνορα και να διευρύνει την εμβέλειά της. Το Ισραήλ δέχτηκε να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα για να αποσταλούν τρόφιμα. Μόνο μια άμεση εκεχηρία όμως θα επιτρέψει τη μαζική μεταφορά τροφίμων που χρειάζεται η Γάζα. Και αυτό αφορά και την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών το Ισραήλ θα πρέπει να επιτρέψει το άνοιγμα των ανθρωπιστικών ε, διαδρόμων για να μεταφερθούν ε, τρόφιμα και ιατρικά είδη καθώς και καύσιμα στον πληθυσμό της Γάζας και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και ένας ελεύθερος διάδρομος διέλευσης σε ολόκληρη την ε, λωρίδα της Γάζας. Αυτή όμως η λύση δεν αρκεί για την ειρήνευση στην περιοχή. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με πιο διευρυμένα, διευρυμένες προκλήσεις, να έχουμε μία ολιστική στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής και να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις που σταμάτησαν εξαιτίας της κρίσης της Γάζας. Πιστεύω ότι για μια ακόμα φορά θα πρέπει να προωθήσουμε τα αιτήματα του Παλαιστινιακού ε, λαού και θεωρούμε ότι η Αιγυπτιακή πρωτοβουλία κινείται προς ε, αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει οποιαδήποτε παλαιστινιακή κυβέρνηση που προωθεί μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις ε, αρχές του κουαρτέτου. Θα πρέπει να αποζητήσουμε μία ε, βιώσιμη και εκτενή ειρηνευτική προσπάθεια στη Μέση Ανατολή και θα πρέπει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης για την επίλυση της ε, σύραξης στην Ευρώπη. Μια βιώσιμη λύση εξαρτάται από την εξέλιξη της ε, κατάστασης στα σύνορα και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να επιτευχθεί η ειρήνη και στις δύο πλευρές, και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη θα πρέπει να έχουμε αναγνωρισμένα και ασφαλή σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μία ειρηνευτική επίλυση το, της σύραξης αυτής, γιατί η πολιτική ζημία είναι πολύ μεγάλη εξαιτίας της πόλωσης και της διεύρυνσης της ε, σύραξης. Ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα οδηγήσει στην ειρήνη στην ε, περιοχή αυτή που έχει πληγεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι προς συμφέρον του ιδίου του Ισραήλ και των γειτόνων του. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή τη βλάβη που έχει επιτελεστεί εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών και τώρα η κυρία Φέρο Βάλτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το κάνω εγώ κύριε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητά μέλη, πράγματι νομίζω ότι όλοι ελπίζαμε ότι το 2009 θα ξεκίναγε καλύτερα. Δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με μια ε, τραγική κρίση στην Γάζα που διαρκεί για τρίτη συνεχή εβδομάδα. Μας ε, προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία το θέμα αυτό, όπως συζητήσαμε χτες στη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με τα μέλη εκείνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του ε, Σαββατοκύριακου. Ε, βεβαίως ε, αναφέρθηκε ήδη ότι ε, κάθε μέρα είναι όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός των τραυματιών και των θυμάτων. Έχουμε και πάρα πολλά άτομα τα οποία υφίστανται εγκάβματα. Οι αρμόδιοι οργανισμοί αναφέρουν ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων πόσο μάλλον η ε, τεράστια αυτή καταστροφή σπιτιών και υποδομής. Όμως και το Ισραήλ είχε απώλειες και ήρθε αντιμέτωπο με εκατοντάδες πυράβολων που εκτοξεύθηκαν στο έδαφος του από τη Χαμάς με στόχο τον άμαχο πληθυσμό. Δυστυχώς όλα αυτά οδηγούν σε να υπάρχει μεγάλη ε, μεγάλος πόνος και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν πέρα από τις ε, καταστροφικές συνέπειες, η κατάσταση αυτή αναβάλει όλο και περισσότερο, μεταθέτει όλο και περισσότερο την προοπτική της ειρήνης, ε, φαλκιδεύει την όλη διαδικασία και θα έχει πολύ ενδικές συνέπειες στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Θα ήθελα σύντομα να σας ε, παρουσιάσω και τις διπλωματικές ενέργειες τις οποίες αναλάβαμε για να πάυσει αυτή η σύραξη και να αντιμετωπίσουμε τις μέσω μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δραστηριοποιηθήκαμε ήδη από την πρώτη μέρα. Δεν ήμασταν οι πρώτοι παίκτες, ήμασταν όμως ένας σημαντικός παίκτης. Και θεωρώ λοιπόν, απαντώντας στο ξέσπασμα της ε, κρίσης, είχαμε την ε, έκτακτη συνάντηση στο Παρίσι των Υπουργών Εξωτερικών στις 30 Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να προετοιμαστούν οι ε, προτάσεις, η δήλωση του Παρισιού και να πάψει αυτή η εξήρα ε, στη Μέση Ανατολή. Έχουμε λοιπόν εδώ τρία βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη δήλωση των Παρισίων που η δήλωση αυτή απαιτεί ε, την ε, κατάπαυση του πυρός, την άμεση κατάφαση του πυρός την ε, πάυση της εκτόξευσης πυράβλων ε, από τη Χαμάς ε, αλλά και την αναστολή όλων των Ισραηλινών ενεργειών. Ζητήσαμε η κατάπαυση του πυρός να σύνοδευθεί από, μια, από, ένα, το άνοιγμα των σημείων διέλευσης κάτι παρεμφερές συνέβη το 2005. Εκφράσαμε την προθυμία μας να επιτρέψουμε το άνοιγμα του σημείου διέλευση στη Ράφα, να μην υπάρχουν πλέον εκεί οι βομβαρδισμοί και να επανεξετάσουμε τη δυνατότητα να χορηγηθεί βοήθεια και σε από άλλα σημεία διέλευση υπό την προπόθεση ότι θα καλυφθούν οι ανησυχίε μα περί ασφαλεία. Βεβαίω και υπογραμμίσαμε τι επίγουσε ανθρωπιστικέ ανάγκε και είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν. Ε, ζητάμε το άμεσο άνοιγμα των σημείων διέλευση για να περάσουν τα φάρμακα, να διανομηθούν τα τρόφιμα στη Γάζα να μπορέσουν οι ε, εργαζόμενοι στο ανθρωπιστικό τομέα να δραστηριοποιηθούν και για να εκενωθούν ορισμένες περιοχές. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε αυτή την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι ο μόνος σωστός τρόπος και οι προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν μόλις επικρατήσει κατάπαυση του πυρός ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ε, θα ακούσατε, τη δική μας την αποστολή την συνδυάσαμε και με την επίσκεψη του κυρίου Σαρκοζή, ο οποίος είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Συρία και το Λίβανο και αποφάσισε να πάει και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο για να ενισχύσει όλες αυτές τις προσπάθειες πάντα με βάση τη δήλωση της 30ης Δεκεμβρίου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς είχαμε ένα πολύ καλό συντονισμό, ε, κοινή συνάντηση στη Ράμα αλλά όπου ο πρόεδρος κ. Ε, Σαρκοζή παρουσίασε το δικό του το πρόγραμμα παύση του πυρό και εμείς η Τρόικα ε, είχαμε επιτόπου προετοιμάσει τις συζητήσεις μας με τις εμπλεκόμενες πλευρές κυρίω με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Ε, στείλαμε λοιπόν ένα ισχυρό ενωτικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα αυτή την ευρωπαϊκή θεσμική θέση κατέστησε σαφές το μήνυμά μας. Αυτό επίσης ε, το παρουσιάσαμε και στον κύριο Σαρκοζή και στον κύριο Σολάνα, ο οποίος ε, πήγε και στη Συρία και στη Λίβανο και ήρθε και σε διαβουλεύει με την Τουρκία. Όλα αυτά ήταν απολύτως απαραίτητα. Εγώ επέμεινα ειδικά στην ανθρωπιστική κατάσταση, <clears throat> όπως ήδη αναφέρθηκε, και ζήτησα ε, επιτακτικά το άνοιγμα των σημείων διέλευση και επίσης και τη δυνατότητα, τουλάχιστον για κάποιες ώρε να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Το Ισραήλ δέχθηκε κάποιο από αυτά τα σημεία και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να υπάρχει σωστός συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας με τη βοήθεια των Ισραηλινών ε, στρατιωτικών δυνάμεων όπως ακριβώς είχε γίνει κατά τη διάρκεια του ε, πολέμου στο Λίβανο. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό μέσα για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους θαραλέους συναδέλφους που εξακολουθούν να δουλεύουν στην Γκάζα, αυτούς από την Άνρα και ε, αυτούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι χρηματοδοτούνται από εμάς αλλά ευχαριστώ και όλες τις άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρωπιστικών ε, ε, λειτουργών που έπεσαν θύματα. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν έχει διαθέσει ήδη σημαντικά κονδύλια για ανθρωπιστική βοήθεια και είμαστε πρόθυμοι να ε, διαθέσουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Όπω είπε ο Προεδρεύων, λοιπόν, το βασικότερο ή τα βασικότερα στοιχεία υπήρχαν ήδη και πριν από την τελευταία ε, δήλωση, ε, το ψήφισμα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας, λίγες μέρες μόνο μετά την έγκριση και την περάτωση των διαπραγματεύσεων, στο ψήφισμα απήχαν οι Αμερικανοί. Η Αίγυπτος εγγυάται να μην υπάρχει λαθρέα μετακίνηση μέσω των σειράγκων, να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη δυνάμεων, ενδεχομένως με διεθνή συμμετοχή και με τη συμμετοχή των ε, σωμάτων ασφαλείας ε, των, ε, της Παλαιστίνης να υπάρχει ένας διάδρομος στη Γάζα. Από ό,τι ξέρουμε η Παλαιστινιακή Αρχή δέχθηκε αυτή την πρόταση και τώρα το Ισραήλ και η Χαμάς μελετούν την πρόταση αυτή και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να γίνει κάτι συντομότατα η τελευταία, σύμφωνα με τι τελευταίες πληροφορίε που έχω, πράγματι όλοι εξετάζουν ενδελεχώ αυτή την πρόταση και ίσως μετά από κάποιες μέρες να έχουμε ε, πάυση πυρό διαρκεία. Εγώ τουλάχιστον ε, το εύχομαι με όλε μου τις δυνάμεις. Τώρα, μέσω πρόθεσμα, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς πρώτα απέρριψαν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, όμως ε, από τις ε, επαφές που είχαμε εικάζω ότι τελικά μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία. Σύντομα, είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αίγυπτος έπαιξε ηγετικό ρόλο στις άμεσες επαφές με τη Χαμάς και βεβαίως ο πρόεδρος κύριος ε, Σαρκοζή με την επίσκεψή του στη Συρία αλλά και οι τουρκικές προσπάθειες ήταν πολύ σημαντικά βήματα. Εξάλλου, η ε, συνάντηση κορυφής ε, των αραβικών κρατών θα μπορούσε να λάβει χώρα στο τέλος της εβδομάδας στο Κατάρ. Αυτές οι έντονες διπλωματικές ενέργειες δείχνουν ότι στηρίζονται όλοι εκείνοι οι παίκτες ε, που έχουν δυνατότητα επαφής με τη Χαμάς έτσι ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη λύση όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα 1860 των Ηνωμένων Εθνών. Μόλις λοιπόν Λοιπόν συμφωνηθεί η πάυση του πυρός θα πρέπει ίσως ε, να σκεφτούμε το πώς ακριβώς μπορούμε να διαμορφώσουμε πιο συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όμως ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν ε, θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό τον αέναο κύκλο οικοδόμησης και αποδόμησης χωρίς να υπάρχει ειρήνη και ε, ίσως ε, θα μπορούσα κάποια στιγμή να ζητήσω και τη δική σας τη βοήθεια να συμβάλλετε και εσείς στις επικοδομητικές προσπάθειες όπως το έκανα και κατά το παρελθόν. Γνωρίζετε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπανκιμούν ε, περιηγείται την περιοχή και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει και εκείνος σε αυτή την τελική επιτυχία που είναι απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε να έχουμε τη βιώσιμη πάυση του πυρός. Εκείνο που πρέπει να πω είναι το εξής. η επίθεση αυτή οδηγεί στο να αποδυναμωθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους Παλαιστινίους και τους ε, Ισραηλινούς. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ποτέ δεν μπορούν να ε, οδηγήσουν σε ε, ειρήνη διαρκείας. Μόνο μέσα από πολιτικές διαβουλεύσεις μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Και ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει τόσο ανάμεσα στους Ισραηλινούς όσο και με τους Παλαιστινίους. Μόλις λοιπόν θα έχουν πάυσει οι εχθροπραξίες, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξαναξεκινήσουν οι και νομίζω ότι εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ε, διμερεί διαπραγματεύσει ευθύ εξ αρχή. Εδώ λοιπόν ε, χαιρετίζω αυτά που είπε η κυρία Κλίντον, τη δέσμευσή τη, στην οποία προέβη εχθέ. Εμείς ε, θα επιμείνουμε τα εμπλεκόμενα μέρη να διαπραγματευτούν επί της ουσίας και η διαδικασία της Ανάπολης να στεφθεί από επιτυχία. Η κρίση αυτή κατέδειξε ότι ε, είναι πιο απαραίτητο από οποτεδήποτε άλλο να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες. Ε, είναι απίθανο η Χαμάς να εξαλειφθεί από αυτή την επιχείρηση κατά πάσα πιθανότητα. Ε, στρατιωτικά θα αποδυναμωθεί μεν, αλλά θα ενισχυθεί πολιτικά η θητεία του ε, κυρίου Αμπάς ε, τελειώνει στις 19 Ιανουαρίου και αυτό επίσης είναι ένα θέμα γιατί έχει σχέση με τη μεταρρυθμίση της PLO και της ΦΑΤΑΧ. Για να επιτευχθεί η ειρήνη διαρκείας είναι σαφές ότι μια ισχυρή Παλαιστινιακή αρχή πρέπει να εκπροσωπεί όλους τους Παλαιστινίους και ε, πρέπει να δεσμεύσουν να υπάρξουν δύο κράτη να συσταθούν αυτά με ειρηνικά μέσα. Η σύγκρουση στη Γάζα δυστυχώς έχει και αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την περιφερειακή στήριξη της ε, διαδικασίας ειρήνης. Έχουμε ε, αραβικά καθεστώτα ε, φιλοειρηνικά τα οποία όμως έχουν εξοργιστεί με την κατάσταση στη Γάζα οι ηγέτες του Ισραήλ αλλά και οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι όλα αυτά είναι πολύ αρνητικά για τις ε, προσπάθειές τους που είναι ίσως να υπάρξει ειρήνη. Εμείς λοιπόν πρέπει να τους πούμε ότι ε, το Ισραήλ δεν μπορεί πλέον να αφήνει να χάνεται χρόνο ε, στη διαδικασία επίτευξης ειρήνης. Αγαπητοί βουλευτές, αυτή είναι η πρώτη μου σύντομη, κάτω μάλλον ή ανάλυση. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να υπάρξει πάυση πυρός διαρκείας και μετά να προχωρήσουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης σε συνεργασία με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Πάμε τώρα ε, στη συζήτηση και στις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος ε, Σαλαφάνκα εκ μέρους του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Δεκαοκτώ ημέρες έχει μέχρι τώρα διαρκέσει η επιχείρηση στη Γάζα με πολλές απώλειες, ιδιαίτερα σκοτωμό αμάχων, χάος, μίσος, αντίδραση και βεβαίως επικράτηση των ριζοσπαστικών στοιχείων έναντι των μετριοπαθών, διότι όπως είπε και ο Προεδρεύων, μπορούμε να κερδίσουμε όλες, όλες τις μάχες σε έναν πόλεμο, αλλά μπορούμε να χάσουμε τη βασικότερη μάχη που είναι η ειρήνη θα πρέπει όχι να επιρρύπτουμε ευθύνες στους μεν ή στους δε, αλλά να φτάσουμε σε μία άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως ορίζει το ψήφισμα 1860 των Ηνωμένων Εθνών και να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα την οποία ελέγχει η Χαμάς που εγγράφεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που οδήγησε σε αυτές τις συνέπειες. Η πολιτική μας ομάδα θα ήθελε να υποστηρίξει την αυριανή πρόταση ψηφίσματος και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπροκ, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει σκληρές διαπραγματεύσεις. Θα θέλαμε σε συνεργασία με άλλα αραβικά κράτη όπως την Αίγυπτο και με τα μέλη του κουαρτέτου να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Επίσης, χαρήκαμε ιδιαίτερα με τις χτεσινές δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον έτσι ώστε να καταβάλουμε μια προσπάθεια επίλυσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών. Η μεγαλύτερη αξία είναι η ειρήνη. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και γι' αυτό ακριβώς θα συνδράμουμε και εμείς. και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ανθρωπιστικές συνέπειες και απόρριες της όλης αυτής τη Κύριος Σούλτς, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. <clears throat> Τέτοιου είδου συζητήσεις όπως ε, οι σημερινοί είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι δύσκολες διότι το Ισραήλ ε, είναι ένα κράτος φιλικό προς εμάς και εγώ προσωπικά ε, μπορώ να το πω αυτό, πολλοί από εμάς ε, αισθάνονται ότι έχουν μια βαθιά φιλία με αυτό το κράτος. Ακόμα σημαντικότερο λοιπόν είναι το ότι θα πρέπει κανείς με τους ε, φίλους να μιλάει ανοιχτά για επίμαχα θέματα. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτή η σύγκρουση οδήγησε σε χίλιους νεκρούς σε 17 ημέρες. Είναι μια πολύ αιματηρή επίθεση και από αυτή την επίθεση υποφέρουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Έχουμε λοιπόν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και με βάση αυτό θα μπορούσε κανείς να διαπραγματευτεί την κατάπαυση του πυρός. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι η σύγκρουση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο ε, το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να ε, τηρούνται. Αυτό λοιπόν είναι κάτι αυτονόητο για ένα δημοκρατικό κράτος και είναι κρίμα που πρέπει να συζητάμε για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η έκκληση να συγγύσουν ε, τα όπλα είναι επιτακτική έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι κάτι το τυχαίο το οποίο αναφέρουμε στο ψηφισμά μας. Είναι ζωτική σημασίας για να αποτρέψουμε τον θάνατο, τον, ε, τους, ε, την πείνα, ε, και τη μιζέρια, τον πόνο, την εξαθλίωση. Υπάρχει βέβαια το δικαίωμα αυτοάμυνας του κράτους του Ισραήλ. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχει το δικαίωμα αυτού του κράτους να υπεραμείνεται απέναντι σε ε, ανθρώπους τρίτους που έχουν στόχο να καταστρέψουν το κράτος αυτό. Όμως ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να διερωτάται πάντα κατά πόσον τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι ανάλογα αυτού που θέλει να πράξει, να επιτύχει. Και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου, όπως και εγώ, πιστεύουν ότι αυτή η αναλογία δεν υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι ανεξάρτητα ε, από ποια πολιτική παράταξη είναι οι φίλοι μας στο Ισραήλ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Χαμάς δεν είναι ειρηνευτικό κίνημα γνωρίζουμε ότι στη Χαμάς ε, το πάνω χέρι το έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμερίζονται τις δικές μας τις ε, αξίες και Βεβαίω, ε, η επίθεση κατά του Ισραήλ οδηγεί στο να πρέπει και το κράτο αυτό να αμυνθεί. Παρόλα αυτά όμω είναι πλάνη το να αρνείται κανεί το διάλογο. Γιατί αν ο διάλογος είναι ε, προϋπόθεση εκ των όνουκάνευ ε, για μια ειρηνική ρύθμιση, το να αρνείται κανείς το διάλογο κατ' ουσίαν αυτό σημαίνει ότι διαιωνίζεται ο ενόπλος αγώνας. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρξει μια ζωτική διόρθωση. Ναι, φοβάμαι πρέπει κανείς να μιλήσει με τη Χαμάς. Αν ε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό απευθείας στο Ισραήλ και αυτό το κατανοώ οι Ισραηλοί πολιτικοί λένε ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ε, μαζί τους ε, παρότι υπάρχουν αρκετοί Ισραηλοί που ε, πιστεύουν ότι πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση. Όταν όμως η κυβέρνηση ή οι βουλευτές του Ισραήλ λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί της, υπάρχουν ε, άλλες δυνατότητες όπως η τετραμερής. Και στο πλαίσιο της τετραμερούς είναι μεταξύ άλλων και η διαμεσολάβηση για να υπάρξει διάλογος. Είναι λοιπόν λάθος να πιστεύει κανείς ότι στο τέλος αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα υπάρξει μια στρατιωτική λύση. Αυτό είναι κεφαλαιόδες ολίσθημα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν θα υπάρξει καμία λύση μέσα από τρομοκρατικές επιθέσεις, ούτε και θα υπάρξει λύση μέσα από συμβατικές στρατιωτικές επιθέσεις. Η μόνη λύση που μπορεί να εξευρεθεί είναι μέσα από τη συμπερίληψη της ε, διεθνούς διαμεσολάβησης. Η πάυση του πυρός ε, είναι επιγόντως απαραίτητη, γι' αυτό λοιπόν ο μηχανισμός που διαθέτει η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινητοποιηθεί με τη ε, συμμετοχή των αραβικών και κυρίως μουσουλμανικών κρατών. Αυτή είναι μια δυνατότητα έτσι ώστε να επιτευχθεί η πάυση του πυρός τώρα και να υπάρξει βελτίωση. Όταν εγώ ήμουν νεαρός και μπήκα στην πολιτική, τότε μου είπανε, ξέρεις, με τους τρομοκράτες δεν μιλάμε τότε ο μεγαλύτερος τρομοκράτης, ξέρετε ποιος ήταν, ο Αραφάτ. Και μετά από κάποια χρόνια είδα στην τηλεόραση αυτός ο τρομοκράτης να παίρνει το βραβείο Νόμπελ μαζί με ε, Ισραηλινούς. Άρα αυτό που δεν είναι δυνατόν τώρα μπορεί να είναι δυνατό στο μέλλον. Έτσι λοιπόν οι μηχανισμοί που υπάρχουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει ο απαραίτητος διάλογος. Εάν λοιπόν το ψήφισμά μας το οποίο ε, εγώ ε, εκ μέρους πολιτικής ομάδας ευχαριστώ για τη σύνταξη του ε, ψηφίσματος. Αν το ψήφισμα αυτό στηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό δείγμα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας. Και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε συμβάλει και εμείς κατά τη μικρή συνεισφορά, αλλά σημαντική για να πάψει να υπάρχει πλέον αυτή η ανυπόφορη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των ε, ε, φιλελευθέρων. Νάιτς Οιτερμπουκ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κάποια μέρα θα πρέπει να πούμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Το πιο κατεπήγον σήμερα όμω, να εκφράσουμε τι απαιτήσει μα να γίνει η κατάπαυση του πυρό, να πάυσει η εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ και να σταματήσουν οι Ισραηλινέ επιχειρήσει στη Γάζα και θα πρέπει να μπορεί να διέλθει ανθρωπιστική βοήθεια μετά μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός να σταματήσει το εμπόριο πυρομαχικών και όπλων με αποτελεσματική επόπτευση των συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, απόσυρση των Ισραηλινών στατευμάτων και εκ νέου άνοιγμα της, των διαφόρων διόδων διελεύσεως άρση του εμπάργκο και όλα αυτά γίνουν ταυτόχρονα. Θα είναι μια φάση περιπλοκότατη που απαιτεί αναμφισβήτητα πιθανότατα την παρουσία διεθνούς δυνάμεως και η Ένωση θα πρέπει να ετοιμαστεί να συμμετάσχει σε αυτήν. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Για να πετύχουμε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει και να δρά σαφώς και όχι κατακαιρματισμένα. Τα καλά συναισθήματα είναι καλά, αλλά σημαντικότερη είναι η αποτελεσματικό της. Θα πρέπει επίσης η ΕΠΑ να συμμετάσχει στις προσπάθειες καθώς και, Ευρωπαϊκός, και ο Αραβικός Σύνδεσμο και τα κράτη-μέλη του Αραβικού Συνδέσμου. Για να προσφερθεί πραγματική εναλλακτική όσον αφορά την κατάσταση Γάζα το Ισραήλ θα πρέπει να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση στην Δυτική Όχθη. 134 σημεία ελέγχου που διακόπτουν τα δίχτυα και τύχη ύψους 8 μέτρων συν ε, διάφορη, μια συμπεριφορά εκνευριστική για τους Παλαιστινίους δεν ε, διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων της Γάζας και δεν ε, βοηθά να απομακρυνθούν από τη Χαμάς. Και τέλος, αναπόφευκτα, θα έρθει η μέρα που όλος ο κόσμος θα πρέπει να μιλήσει με όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, τη Ευρώπη ε, των Εθνών, κυρία Μουσκαρντίνη. Κύριε Πρόεδρε, όπω όλοι, προφανώ ε, έχουμε ταραχθεί από αυτήν την κατάσταση και συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, όμω υπάρχει καθήκον τουλάχιστον από την πλευρά μου, πιστεύω, να καταγγείλουμε οποιαδήποτε υποκρισία Λοιπόν, ε, ξεκινάμε πολύ μακριά ιστορία. Είναι το δικαίωμα το καθαγιασμένο των Παλαιστινίων να έχουν μια χώρα ελεύθερη, ένα κράτος ελεύθερο και περνά από το επίσης ιερό δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να αναγνωρίζεται. Και γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ ακυρώθηκε από το γεωγραφικό χάρτη, διαγράφει από το γεωγραφικό χάρτη πολλών χωρών. Ε, γνωρίζουμε ότι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, σίγουρα δεν θα είχαν ανεχθεί να έχουν διαγραφεί από το γεωγραφικό χάρτη. Δεν θα είχαν δεχτεί να θεωρούνται σαν ανύπαρκτες χώρες. Και ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Είναι η τρομοκρατία βασικός, βασικό αίτιο, βασικό πρόβλημα. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι άνευ υποκρισίας σήμερα έχουμε καθήκον να ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα θέμα διαφορετικά. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι ο διάλογος με τους τρομοκράτες δικαιολογείται από το γεγονός ότι πέθαναν τόσοι πολίτες άμαχοι, διότι αυτό δημιουργεί δικαιολογία για οποιοδήποτε μελλοντικό τρομοκράτη να χρησιμοποιεί τη βία, την ισχύ και το θάνατο για να πετυχαίνει την νομιμότητα την πολιτική. Πιστεύω ότι θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να βρούμε μεγαλύτερη συνοχή, τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε και τις οικονομικές σχέσεις με τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ, να αγγιηθούμε διόδους για ανθρωπιστική βοήθεια, ούτω ώστε οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί άμαχοι πολίτε να μπορεί να είναι ασφαλεί σε αυτή την περίπτωση. Περισσότερο αυτό αφορά του Παλαιστινίου που υποφέρουν. Και τούτου λεχθέντος κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι θα ήταν καλό και σκόπιμο να επανεξεταστεί αυτή η θέση που έχουμε όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούμε και δεν ελέγχουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση ε, σίγουρα είναι φρικτή ελπίδα ειρήνης και ασφαλείας για τους μεν και τους δε εξατμίζεται στους καπνούς της Γάζας και κάτω από τα σώματα των νεκρών, των παιδιών και των γυναικών και των ανδρών και των πληγωμένων. Απέχουμε πολύ από την ελπίδα για ασφάλεια, περισσότερο μακριά τώρα από ποτέ. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτός ο πόλεμος εντάσσεται στη λογική της Ισραηλινή επιχειρηματολογία, ένας πόλεμο που δικαιολογείται από το γεγονός ότι υπήρξε επίθεση με ρουκετών που εκτοξεύονται κατά του Ισραήλ ότι αυτό δικαιολογεί να δοθεί ένα μάθημα στους Παλαιστινίους δεν έχω καταλάβει τίποτα, τίποτα δεν κατάλαβαν διότι το να δώσει κανείς ένα μάθημα είναι μαύρη παιδαγωγική, ποτέ δεν λειτουργήσε από τον Κλαούζεβιτ. Ξέρουμε ότι αυτό που ξεκινά έναν πόλεμο πρέπει να ξέρει πώ να το σταματήσει. Πρέπει να ξέρει ποιο είναι ο στόχο. Και ο στόχο αυτού του πολέμου είναι περισσότερη ασφάλεια για το Ισραήλ. Και μπορούμε να πούμε ήδη από σήμερα ότι ο στόχο αυτού του πολέμου δεν θα είναι ποτέ εφικτό μέσω αυτού του πολέμου και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτό ο πόλεμο. Όσο περισσότερο σκοτώνει κανεί αμάχου πολίτε, όσο σκοτώνει Παλαιστινίου, λιγότερη ασφάλεια θα υπάρχει στην περιοχή. Αυτό είναι το δράμα. Αυτή είναι η τραγωδία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή την περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Ο Μάρτιν Σούλτ έχει δίκιο θα πρέπει να προστατεύσουμε το Ισραήλ έναντι του Ισραήλ. Να προστατεύσουμε το Ισραήλ από τον πειρασμό να βρει τη λύση του πολέμου και τη λύση του στρατού. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, Παλαιστινίους έναντι της Αμάς. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, Παλαιστίνιους πολίτες απέναντι στη Χαμάς. Ιδού. Αυτό είναι το καθήκον μας, το έργο μας. Δεν είναι εύκολο αλλά θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ε, ζητώ από το Συμβούλιο να σταματήσει να εξετάζει το upgrading, τη βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ, όσο η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Είναι κακή λύση. Δεν είναι η καλή λύση. Ζητώ, ζητώ από όλους εκείνους οι οποίοι σωστά προτείνουν διάλογο, συζήτηση με τη Χαμάς, να μην είναι αφελείς να έχουν στο κεφάλι τους ότι πρέπει να συζητήσουν με την Χαμάς για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Γάζα εφόσον έχουν την εξουσία. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουν ότι η Χαμάς ε, χρειάζεται τους θανάτους για να ζει. Και το Ισραήλ έπεσε στην παγία της Χαμάς. Όσο υπάρχουν νεκροί στη Γάζα, καλύτερα είναι για τη Χαμάς. Ιδού λοιπόν μία από τις αλήθειες που θα πρέπει να πούμε στη Χαμάς. Αρνούμεθα αυτή τη στρατηγική, την αυτοκτονική της Χαμάς η οποία θέλει να δημιουργεί θύματα και μάρτυρες για να ε, επιτεθεί κατά του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να το πούμε στη Χαμάς επίσης. Για να κλείσω θα πω ένα πράγμα. Οι μόνοι που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της Χαμάς είναι οι Παλαιστίνοι. Εφόσον το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείπει την κατοχή της Δυτικής Όχθης, Όσο το Ισραήλ δεν θα δώσει μια λύση θετική στους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης, όλο και περισσότερο οι Παλαιστίνοι θα πάνε και θα στραφούν προς την Χαμάς. Αν δώσουμε μια ελπίδα ζωής στη δυτική όχθη στους Παλαιστινίους, οι Παλαιστίνοι θα επαναστατήσουν κατά της Χαμάς και θα μας απαλλάξουν από την Χαμάς. Θα απαλλάξουμε τους Παλαιστινίους από την κατοχή του Ισραήλ στη δυτική όχθη και οι Παλαιστίνοι θα απελευθερωθούν από την Χαμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρου τη Ενωμένη Αριστερά. Η κυρία Μοργαντίνη, δυόμιση λεπτά. Ένας Παλαιστίνιος έχασε τα, τα παιδιά του, το σπίτι του και συγγενεί. Και μας είπε με μεγάλο άγχος ότι η Χαμάς θα πει ότι νίκησε όταν σταματήσει αυτή η επίθεση. Το ίδιο θα πει και το Ισραήλ. Στην ουσία όμως χανόμαστε εμείς οι άμαχοι. Και βλέπουμε αυτά τα πτώματα των αμάχων, των γυναικών, των παιδιών. Οι τραυματίες που είναι 4.000 βρίσκονται στα νοσοκομεία και δεν τους παρέχονται βοήθειες. Εδώ πεθαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία καταπατώνται και αυτή είναι μια τραγωδία. Εμείς είμαστε αναποτελεσματικοί. Κυρία ε, Μπενίτα Φερεροβάλνερ, ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερα και ξέρω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε μαζί με άλλους. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε σαφέστατα ότι αυτός ο στρατιωτικός νόμος και πόλεμος δεν σώζει το Ισραήλ. Και όπως είπε ο David Grossman, όταν σκοτώθηκε ένας ραβίνος, σκοτώθηκε γιατί υποτίθεται ότι ήθελε να προωθήσει την ειρήνη. Ας ε, σταματήσετε, ας καταπέσετε πάψετε το πυρ. Υπάρχει ε, ένας Νορβηγός εκπρόσωπος μίας ε, μη κυβερνητική που μας λέει τι συμβαίνει. Μιλάμε για διπλωματία, αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο τη διπλωματία, αλλά όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Ένα από αυτά και για το Ισραήλ αφορά το upgrading τη βελτίωση των σχέσεων και χαίρομαι διότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τελαβίβ είπε ότι ας μην μιλάμε για upgrading, ας ε, σταματήσουμε για λίγο ότι αυτό που έχει σημασία είναι η κατάπαυση του πυρός επί του παρόντος. Μας μιλούσε λοιπόν για διεθνή προστασία. Δεν σκεφτόμαστε μόνο τη Γάζα και τη Ράφα. Μιλάμε για προστασία για τους άμαχους που έρχεται από το βορρά από τις ε, Ισραηλινές επιθέσεις από το βορρά. Ο έλεγχος των σειρώνων είναι γενικός από τον νότο, από τη Ράφα μέχρι το βορρά. Γιατί μετά το 1992 από τη Συμφωνία του Όσλο οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να βγουν από τα σύνορα του βορρά και να πάνε στο νότο στη Ράφα. Ξέρετε λοιπόν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τούνελ, να εξοπλίσουν την ΑΜΑΣ, αλλά δεν έχουν ελεύθερη διέλευση. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε όλα τα σημεία διέλευσης. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν τρόφιμα, εάν δεν έχουν εμπόριο, τότε θα πρέπει να ασκηθεί πίεση έτσι ώστε η Χαμάς να μην προωθεί αυτή τη δράση, αλλά υπάρχει και η δυτική όχθη και δεν θα πρέπει να γίνονται άλλοι ούτε επικισμοί ούτε επιθέτηση. Ευχαριστούμε την Λουίζα Μοργαντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοργαντίνη. Πραγματικά υποκλίνομαι σε εσά ε, για το γεγονός ότι από κοινού με του συναδέλφους επισκεφθήκατε επιτόπου τη λωρίδα της Γάζας. Επόμενος ομιλητής ε, από τους ανεξάρτητους ε, για ένα λεπτό κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Παλαιστίνη είναι Ισλαμικό, Ισλαμική περιοχή και Ισλαμικό κίνημα η Χαμάς βασίστηκε σε αυτή την αρχή. Υποστηρίζεται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν η Χαμάς. Αν το δει κανείς από αυτή την ιδεολογική σκοπιά, δεν υπάρχει χώρος για το κράτος του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες του μουσουλμανικού ολοκληρωτισμού αυτού είναι η ματιρία αυτή σύραξη στην λωρίδα της Γάζας. Όσον αφορά τη Χαμάς λοιπόν, η Χαμάς ωφελείται από τον πόλεμο αυτό. Αν η Ευρώπη πραγματικά επιθυμεί να εξασφαλίσει τη διαβίωση του κράτους, την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ, τότε θα υπάρξει αντιπαράθεση με την Χαμάς. Αυτή η προοπτική χρειάζεται σωστή προετοιμασία, διότι η κατάπαυση του πυρός είναι απλώς ένα διάλειμμα για την Χαμάς εάν συμφωνήσει με μια κατάπαυση του πυρός. Δεν θα είναι μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ο κ. Ρωμανιόλη, 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου συμμερίζεται τις ευχές για την ειρήνη και τις ανησυχίες που μέχρι τώρα εξεφράστησαν από πολλούς. Πιστεύω και όσα υποστηρίχθηκαν από το Συμβούλιο μπορούν να μα βρίσκουν συμφώνους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε μια δρομή που είναι χρήσιμη για το διάλογο. Άνοιγμα των διαλέψεων για ανθρωπιστική βοήθεια, κατάποση του πυρός διμερής ίσως να είναι και πρόδρομος για μια διοργάνωση ε, μέσω διεθνού δυνάμεως. Έχει δίκιο η κυρία Μοργαντίνη, συνάδελφο Μοργαντίνη που ζητά αυτή η λύση, αυτή η διέλευση, αυτή η λύση να αφορά όλο το παλαιστινιακό πρόβλημα. Ε, η κυρία Φερέρο Βάλτνερ ε, εύχεται να συνεχιστούν διπλωματικές διεργασίες. Ίσως μπορούμε να ακολουθήσουμε και αυτά που είπε και ο Πάπας. Πρέπει να προσπαθήσουμε μετά από πολλά χρόνια να βρούμε μια λύση για δύο λαούς, δύο κράτη. Δεν πρέπει να το λησμονούμε και επιτέλους πρέπει να επιβεβαιωθεί, το, να απαγιωθεί το διεθνές δίκαιο. Δεν θα υπάρξει ποτέ λύσεις καλή, όπως είπε ο κύριος Σούλτς, πρέπει να το επιθυμίζω που και που και αυτόν, μια λύση ποτέ δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν βρεθεί ε, κάποια λύση για τα περιοχή των Αγίων Χωμάτων. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε διπλωματική προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Ο συνάδελφο κύριος ε, Σούλτ, ε, φαντάζομαι θα χάλει και πάρα πολύ που ε, τον αναφέρατε από κοινού με τον Άγιο Πατέρα. Ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Κύριε, βλέπω και τον κύριο Σούλτ μπροστά μου. Λοιπόν, να πω το εξή: Έχουμε τη Χαμάς η οποία είναι κατά της λύσης των δύο κρατών η οποία απορρίπτει το δικαίωμα του Ισραήλ ε, να υπάρχει, η οποία ε, πραξικοπηματικά επέβαλε κάποιους ανθρώπους με ρουκέτες, ε, βάλει κατά το, το αμάχου πληθυσμού και χρησιμοποιεί ανθρώπους ως ανθρώπινη ασπίδα. Τι θα πρέπει λοιπόν τώρα να γίνει, πώς θα πρέπει κανείς να αντιδράσει τη στιγμή που η ίδια η Χαμάς χρησιμοποιεί ανθρώπους για ανθρώπινη ασπίδα. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα της αναλογικότητας, το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί σε αυτή την περίπτωση. Σε πόλεμο δεν υπάρχει αναλογικότητα, όλοι οι πόλεμοι και ο ένας νεκρός είναι παραπάνω από ό,τι θα πρέπει να υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι η βασική αρχή. Γι' αυτό λοιπόν δεν ε, θα πρέπει να αποδίδουμε ενοχές ή ευθύνες, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και θεωρώ ότι ο κύριος Φάτσεμπερκ με την αντιπροσωπεία του και η Επίτροπος η κυρία Φεραρο Βάλτνα και με τη βοήθεια άλλων εθνικών αντιπροσωπιών έκαναν πολλά περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Ούτε τους Αμερικανούς είδα, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε μέλη του ε, κουαρτέτου παρά μόνο αυτούς που σα ανέφερα. Γι' αυτό και του ευχαριστούμε. Και ω εκ τούτου η κατάπαυση του φυρός πρέπει να περιλαμβάνει το κινήσει από πλευράς του Ισραήλ αλλά και κινήσεις από πλευράς της Χαμάς τις ρουκέτες που έχει από την Κορέα και το Ιράν να μην τις εκτοξεύει κατά του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησει μέσα από διεθνείς συμφωνίες συμπεριλαμβανομένου και της, συμπεριλαμβανομένης της τετραμερούς και της Αιγύπτου να υπάρχει τέτοιο έλεγχο των συνών έτσι ώστε οι ρουκέτες να μην μπορούν να περάσουν. Και τέλος ε, θα πρέπει να πάυσει αυτή η Ισραηλινή επίθεση. Κυρίες και κύριοι, μία τελευταία μου παρατήρηση. Αυτό είναι το πρώτο μικρό βήμα. Στο μέλλον το Ισραήλ αν θέλει να έχει σε Παλαιστινίους αυτό σημαίνει δύο κράτη και επιτέλους θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε οι μετριοπαθείς Παλαιστίνοι και ο πρόεδρος κύριος Αμπάς να μπορούν να επιδείξουν επιτυχίες, να παρουσιάσουν τις επιτυχίες αυτές στους πολίτες. Να μην υπάρχει πια επικιστική πολιτική, γιατί αν δεν υπάρχουν επιτυχίες κερδίζουν όπως καταλαβαίνετε οι ακραίοι και νομίζω ότι εκεί έγκυται η λύση του ε, προβλήματος. Ε, πρέπει να πω ότι δεν χρησιμοποιήσετε καλά το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Η κυρία Ναπολιτάνο. Μιλάμε για μια μεγάλη τραγωδία, άρα τα λόγια μας είναι ανεπαρκή. Έχουμε να κάνουμε με ένα στρατό που σκοτώνει εκατοντάδες ε, χιλιάδες ανθρώπους και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο της τρομοκρατίας που υποτίθεται θέλει να κατατροπώσει. Όποιος γνωρίζει τη Γάζα και αν τη δει στο χάρτη και μόνο, ξέρει ότι καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να οργανωθεί χωρίς να λάβει υπόψη την θανάτωση αμάχων. Το Ισραήλ μιλά για μεγαλύτερη ασφάλεια τη στιγμή που δημιουργεί απόγνωση και ποιος θα προσπαθεί να βρει μία οδό διαφυγής σε αυτή την ομιβία, η Χαμάς, Μιλάμε για κατάπαυση του πυρός, όπως ζήτησε και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα θέλαμε να την ε, τηρήσουν οι δύο πλευρές και τα Ηνωμένα Έθνη να την καταστήσουν δυνατή. Αυτή η σφαγή δεν ε, δυνατίζει την Χαμάς, αλλά την Παλαιστινιακή Αρχή. Και εκείνων όσων θέλουν τη διαπραγμάτευση με το Ισραήλ. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ειλικρινά τι έλαβαν υπόψη μέχρι του δε τίποτα. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε εάν θέλουμε πραγματικά να προσπαθήσουμε να κρυζώσουμε το μίσος και τη βία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Ναπολιτάνο και για το γεγονό ότι δεν εξαντλήσετε το χρόνο που έχει προβληθεί για κύριος, Η κυρία Ντεσάρνε για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε και εμεί ένα μερίδιο ευθύνη για όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή. Εμεί, η Ευρώπη και εμεί, η διεθνή κοινότητε. Έχουμε αφήσει να επιδεινωθεί κατάσταση. Αφήσαμε να. δεν κάναμε τίποτα να επιλύτω η ασφάλεια του Ισραήλ και επίσης όταν ε, έγινε το μπλοκάρισμα των, το μπλόκο και έγινε δύσκολη ζωή των Παλαιστινίων. 995 ε, νεκροί έχουμε, 292 παιδιά, χιλιάδες ε, τραυματίες που μερικοί ακόμα περιμένουν να γενοθούν. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που δεν έχουν σπίτι και δεν ξέρουν πού να πάνε. Είναι μια κατάσταση ανθρωπιστική που όλο και χειροτερεύει. 700.000 ε, ε, Παλαιστίνοι τη Γάζα δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό, άλλοι δεν έχουν νερό. Και τρει εβδομάδες διαρκεί αυτό, τρει εβδομάδε όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι ή προσπαθούν να επιβιώσουν μάλλον. Υπάρχει μεγάλο μαρτύριο, μεγάλη δυστυχία, υποφέρουν. Πρέπει αυτό να πάψει, πρέπει να σταματήσει τώρα. Και δική μα ευθύνη εμάς των Ευρωπαίων είναι να μην είμαστε ανεκτικοί εναντί ενός. Ευθύνη ημών των, ημών των Ευρωπαίων είναι να πιέσουμε και τα δύο μέρη τους, ώστε να αποδεχτούν επιτέλους να διαπραγματευτούν. Και είναι ένα θέμα ημερών, ίσως και ωρών, πριν ε, τελικά διαπραχθεί το ανεπανόρθωτο τη χεσέ επίθεση, κυρίω κατά τη πόλη τη Γάζα. Θα πρέπει να εγγυηθούμε στο Ισραήλ την ασφάλειά του. Θα πρέπει να εγγυηθούμε στο λαό τη Γάζα ότι θα μπορεί να ζει αύριο ειρηνικά. Θα πρέπει να ελεγχθούν τα σύνορα και να αρθεί το αποκλεισμό. Όλα, όλοι θα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το, τη συμφωνία. Ίσως θα αρκούσε η Ευρώπη, η ΕΠΑ και οι αραβικές χώρες που θα συνεδριάσουν αύριο να μιλήσουν όλοι μαζί με μία ίδια φωνή, κοινή φωνή. Και να σας πω ποια είναι η πεποίθησή μου, ενδόμηχη σκέψη μου. Ε, δεν είναι ο πόλεμος που θα, θα κερδίσει σήμερα, είναι η ειρήνη που θα πρέπει να κερδίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρομπέρτα Αντζελίλη για ένα λεπτό. Ε, Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους λόγους ε, της Επιτρόπου και του Πρόεδρου Πέτερινγκ που κατήγγυλαν την μεγάλη ευθύνη της Χαμάς σε σχέση με την τήρηση της ε, κεχηρίας. Αλλά νομίζω ότι η αντίδραση δεν είναι αναλογική. Η κρίση παραμένει και υπάρχουν χιλιάδες πολίτες, γυναίκες, παιδιά που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Χωρίς καμία υποκρισία λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε τη στιγμή που τα δικά μας παιδιά γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, πόσα παιδιά πέθαναν στη Γάζα, 200, 300 και πόσοι Ισραηλινοί πολίτες. Πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να κάνει κάτι, κάτι περισσότερο, πολύ περισσότερο, να κατανοήσουμε το βάρος της ευθύνης μας. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε την Χαμάς, να πούμε ποιοι φέρουν ευθύνη, ποιοι περισσότεροι, ποιοι λιγότεροι, αλλά υπάρχει καταρχήν η ανεπάρκεια της Ευρώπης. Μεγάλη ανεπάρκεια και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε μία βιώσιμη στρατηγική ειρήνης. Εμείς σήμερα θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την κατάπαυση του πυρός. Δεν αρκεί αυτό όμως. Θα πρέπει να ορίσουμε όρους συνοδευτικούς της ε, ειρηνευτικής διαδικασίας. Ήθελα να θυμίσω τα λόγια του Πάπα, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να δώσουμε απτές απαντήσεις, έτσι ώστε αυτοί οι λαοί να ζουν σε ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, όπως είπε και η κυρία Μοργαντίνη. Η βία και η φτώχεια είναι οι μεγαλύτερες μάστιγες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μιλήσατε διπλάσιο χρόνο από ό,τι προβλεφθεί για εσάς. Κοιτάξτε, στη Γάζα είδαμε τον πόλεμο, το θάνατο, αλλά είδαμε και νέου ανθρώπου, ανθρώπου που έχουν δικαίωμα να ζουν και έχουμε καθήκον να του προστατεύσουμε. Η προστασία του πληθυσμού των αμάχων είναι κατεπίγουσα ανάγκη, απόλυτη ανάγκη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογεί να μην γίνουν τα πάντα, ούτω ώστε να προστατευτεί αυτό ο πληθυσμό. Και σα το ζητώ, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, σα ερωτώ, έχετε το συνέστημα σήμερα ότι κάνατε τα πάντα, ούτω ώστε να πετύχετε από τι ελληνικέ αρχέ την άμεση κατάπαυση των επιχειρήσεων που αδιάκριτα και δυσανάλογα εκτελούνται, σίγουρα όχι. Ακούμ, όταν οι θόρυβοι, ακούγονταν οι φήμε για τι επιχειρήσει τη πρεσβείας, το Συμβούλιο κατά του Κοινοβουλίου εξέφραζε την απόφασή του να αναβαθμίσει τη σχέση με το Ισραήλ. Ήταν τραγικό σφάλμα. Όταν οι κυβερνητικέ οργανώσει ζητούσαν από το Συμβούλιο Ασφαλεία να, να ζητήσει από το Εθνέ Ποινικό Δικαστήριο να εξετάσει την περίπτωση εγκλημάτων πολέμου, το Συμβούλιο ήταν ανίκανο να κινητοποιήσει τη ρήτρα δικαιωμάτων του ανθρώπου συμφωνία με το Ισραήλ. Βαρέθηκα να ακούω ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε στι προσπάθειε μας. Είναι το αδιέξοδο της πολιτικής σας ουσιαστικά, της ανθρωπιστικής, για να απαλύνετε τις ζημιές της στρατιωτικής κατοχής και του πολέμου, που είναι στο, το μέγιστο της αποτυχίας. Μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε όσον αφορά παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, για να εφαρμόσουμε τελικά τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν δεν είμαστε ικανοί σήμερα να εξετάσουμε την εμβέλεια των αποτελεσματικών μηχανισμών ασκήσεως πιέσεως που πρέπει να εφαρμοστούν, δεν ξέρω πραγματικά ποια κατάσταση θα δικαιολογήσει επιτέλους να κινηθούμε. Και σας το λέω ξεκάθαρα, εάν το business as usual συνεχίσει στη σχέση με το Ισραήλ, θα θάψετε μαζί με τους κύριους νεκρούς της Γάζας το άρθρο 11 της συνθήκης. Θα θάψετε την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ένωσης και θα θάψετε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα ήθελα να παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο σας, ο κύριος Τριντεφυλλίδης, για δυόμιση λεπτά. Επιστρέφοντας από τη λωρίδα της Γάζας, ε, έχοντας δει τη σφαγή κυρίων Σαμάχων, ε, αισθάνομαι ότι πρέπει να εκφράσω την απόλυτη αλληλεγγύη μου με τον Παλαιστινιακό λαό. Για 17 ημέρες αντιμετωπίζουν αυτή την τρομακτική πολεμική μηχανή του Ισραήλ που κατάφορα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Εξάλλου εκφράζω την υποστήριξή μου στις ειρηνευτικές δυνάμεις του Ισραήλ που ζητούν την ε, αναστολή του πολέμου. Μετά από ε, την ε, ε, Τουρκία της Γάζας είδαμε ότι επεκτάθηκαν οι επικισμοί, είδαμε ότι οι δυνάμεις κατοχής μεταφέρθηκαν και εξαπέλυσαν πραγματική επίθεση. Οι ρουκέτες ε, κατά του Ισραήλ και εδώ υπογραμμίζω ότι εγώ είμαι κατά οποιασδήποτε μορφής επίθεσης ε, εις ε, βάρος άμαχου πληθυσμού. Αυτά χρησιμεύσαν ως πρόφαση. Έχουμε ε, και το επιχείρημα ε, δήθεν των εκλογών στο Ισραήλ. Το Συμβούλιο Ασφαλής των Εθνών ενέκρινε ένα ψήφισμα. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος, δεν είναι οργάνωση, είναι μέλος ε, των Εθνών. Έχει την ευθύνη απέναντι στη διεθνή κοινότητα και πρέπει να σέβεται το ψήφισμα αυτό αλλά και όλα τα άλλα τα οποία έχουν εγκριθεί από τα Έθνη. Πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να υπάρχει ατιμορρησία πλέον. Πρέπει να υπάρξουν ολοκληρωμένες διεθνείς έρευνες η διεθνής κοινότητα ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων, ε, την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ελεύθερη μετακίνηση των ε, πολιτών. Ας αφήσουμε τις ειρηνευτικέ δυνάμεις να αναπτυχθούν. Ε, πράγματι, τι κάναμε κάποια βήματα, αλλά μόνο ανθρωπιστικής φύσεως, όχι πολιτικά. Θα πρέπει να ζητήσουμε την αναστολή των, της συμφωνίας σύνδεσης. Να μην υπάρχει βάθμινο σχέση με το Ισραήλ, να μην υπάρχουν όπλα που να εξάγονται στο Ισραήλ, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει υπάρχει άλλη λύση ε, σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να επανέλθουμε στο διεθνέ δίκαιο που σημαίνει ότι πρέπει να πάψει αυτή η κατοχή των 42 ετών τη Παλαιστίνης. Να υπάρχει ένα κυρίαρχο και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτο και με τον τρόπο αυτό να υπάρχει ένα ειρηνικό μέλλον τόσο για τα παιδιά των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών. Για να σώσουμε όμω το μέλλον κύριε Πρόεδρε και τι μελλοντικέ γενιέ, πρέπει τώρα να σταματήσει ο πόλεμο. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο ε, Πάτρικ ε, Λουί, για ένα λεπτό. Εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια ο Δαβίδ ε, αντιμετώπισε το Γολιάθι για να δει κατά πόσο η γη ανήκει στους Φιλιστέους ή όχι. Αυτό ήταν ένας από τους πυλώνες του πολιτισμού μας. Σήμερα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρη ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος το οποίο να είναι κυρίαρχο. Πέρα από τα, τις πολυπολιτισμικές ε, τάσεις υπάρχουν όρια. Εκεί που υπάρχουν δύο λαοί θα πρέπει να υπάρχουν και δύο κράτη με ένα στόχο να προωθήσουμε αυτό το κράτος δικαίου και για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εξτρεμιστές διότι οι μικροί είναι τα θύματα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο στρατιωτικός νόμος δεν μπορεί να ισχύει και οι στρατιωτικές δυνάμεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα πολιτικά. Άλιστερ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η τρομοκρατία είναι κάτι που με κάνει να φρύτω. Η προπαγάνδα της τρομοκρατίας είναι κάτι που αποτάσω. Επειδή είμαι από τη Βόρεια Ιρλανδία, ίσως γι' αυτό είμαι πιο ευαίσθητος. Λοιπόν, όταν ακούω τη Χαμάς να βελάζει ε, όταν μετά από την ε, εκτόξευση πολλών ρουκετών κατά αθών πολιτών κατά του Ισραήλ, τότε δεν εντυπωσιάζομαι, διότι ξέρω ότι η Χαμάς, όπως και ο IRA στη χώρα μου, είναι πολύ καλή όσον αφορά την τρομοκρατία, δάσκαλη όσον αφορά την τρομοκρατία και την προπαγάνδα. Η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Το Ισραήλ δέχεται τη λύση των δύο κρατών. Η Χαμάς δεν μπορεί καν να δεχθεί το δικαίωμα υπάρξεως του Ισραήλ. Έτσι, αένα ε, επιτίθεται τρομοκρατικά και μετά όταν μετά από μεγάλη ανοχή ε, αντεπιτίθεται το Ισραήλ, το παίζει Χαμάς θύμα. Αυτοί είναι που βιοπραγούν. Και αν θέλουν ειρήνη, η απάντηση είναι στα χέρια τους. Σταματήστε να βομβαρδίζετε το Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι κοινή διαπίστωση ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι τραγική αγγίζει τα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. θέλω να συγχαρώ την ευρωπαϊκή επιτροπή για τις ενισχυμένες προσπάθειές της την προεδρία για τις πρωτοβουλίες της και τον συντονισμό της εθνικής κινητικότητας ε, που υπάρχει στον τομέα αυτό καθώς και την αίγυπτο για το σημαντικό και ευαίσθητο ρόλο που παίζει. τώρα είναι επίγουσα ανάγκη η κατάπαυση του πυρός και των εχθροπραξιών από τις δύο πλευρές η διέλευση από τα ισραηλινά εδάφη και από την αίγυπτο για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρωπιστικών και ο έλεγχος των συνόρων για την πάυση της διακίνησης παράνομου πλεισμού και ανθρώπων. είναι θετικές οι ενδείξει, όπως είπε η επίτροπος για ένα σχέδιο εκεχηρία και ελπίζω να γίνει άμεσα δεκτό και σεβαστό στην εφαρμογή του ποια είναι όμως τα επόμενά μας βήματα ήδη έχουν αναφερθεί και από την επίτροπο και από τον προεδρεύοντα του συμβουλίου ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους στόχους μας για την βιώσιμη ειρήνη και τη δημιουργία δύο κρατών ε, ε, ε, ενό παλαιστινιακού κράτου που θα ζει με ειρήνη και σεβασμό δίπλα στο ισραήλ. αυτά δεν είναι καινούρια τα έχουμε διακηρύξει τα έχουμε υποστηρίξει χωρί αποτελέσματα με αρνητικέ συνέπειες ένα φαύλο κύκλο βία και συνέπειε αρνητικέ, όχι μόνο για το λαό του ισραήλ και του Παλαιστινίου, αλλά για όλου του λαού τη περιοχή και για την ασφάλεια τη διεθνού κοινότητα πρέπει τώρα να κάνουμε τον απολογισμό των δράσεών μας των πολιτικών μας επιλογών των πρακτικών μας και να κάνουμε βήματα πιο θαραλέα και διαφορετικά. σε διμερές επίπεδο με το ισραήλ είναι ανάγκη επιτακτική να έχουμε ένα διάλογο ειλικρινή βαθύ μια αυτοκριτική στο πλαίσιο της εταιρικής και φιλικής μας σχέσης για να εντοπίσουμε τα λάθη που έγιναν στην ε, προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών και επίσης να ενισχύσουμε ένα τέτοιο διάλογο με όλους τους παλαιστινίους να τους κάνουμε να καταλάβουν τη σημασία που έχει η ειρήνη η συνοχή η ανθρώπινη ζωή και η ενότητα μεταξύ τους. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σφόμποντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Τοπολάνεκ σήμερα το πρωί έκανε κάποιες ε, αστείες παρατηρήσεις και πρέπει να σας πω ότι εγώ ως Αυστριακός ε, βουλευτής χαίρομαι πάρα πολύ που τόσο η Προεδρία όσο και η Επιτροπή εκπροσωπούνται με Αυστριακούς, από Αυστριακούς. Γνωρίζω βέβαια ότι είστε πιστοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, ε, λίγο πριν από την απόσυρση από τη Γάζα, τότε ο ε, αναπληκτής πρωθυπουργός και πει μην ανακατεύετε θα πάνε όλα μια χαρά. Άλλοι πάλι όπως ε, ο πρώην υπουργό εξωτερικών είχε πει ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν στο χάος. Και πράγματι αυτό συνέβη. το να υπάρχει απόσυρση χωρίς διαπραγματεύσεις αυτό δεν έχει νόημα και εμείς νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να έρθουμε σε επαφή ούτε καν με τους μετριοπαθείς εκπροσώπους ε, της Χαμάς που δεν είναι καν Χαμάς, απλά ορίστηκαν από τη Χαμάς. Δεν είναι σωστό να έρθουμε σε συζήτηση μαζί τους, αλλά το κάναμε, το κάναμε στο παρελθόν και έτσι καταστράφηκε αυτή η ενωτική ε, κυβέρνηση. Ξέρω ότι μερικοί ήθελαν να μιλήσουν αλλά δεν τους επιτρεπόταν Πρέπει λοιπόν να μιλάει κανείς. Ε, η Χαμάς είναι τρομοκρατική εγκληματική οργάνωση και έχει και ε, ζηλωτικές απόψεις. Το θέμα όμως δεν είναι αν χωνεύει δεν χωνεύει κανεί τη Χαμάς. Το θέμα είναι να βρει μια λύση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επανέλθουμε στο διάλογο, ε, κάτι το οποίο είπαν πολλοί συνάδελφοι σήμερα. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα οι άνθρωποι στη Γάζα να μπορούν να ζήσουν μια κατά το μάλλον τον αξιοπρεπή ε, ζωή. Ξέρετε γιατί πάνε στη Χαμάς. Γιατί αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να επιβιώσουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει πρέπει στους ανθρώπους αυτούς να δώσουμε μια οικονομική βάση ε, επιβίωσης. Να μην υπάρχει πια εμπάργο, ούτε μποϊκοντάζ. Και η τελευταία μου παρατήρηση ο συνάδελφος κύριος Μπροκ που τον εκτιμώ είπε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την αρχή της αναλογικότητας και εδώ δεν ερχεί. Ισχύει όμως στο ιδιωτικό δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο ισχύει αυτή η αρχή της αναλογικότητας και όποιος δεν την τηρεί παραβιάζει αυτόματα και το διεθνές δίκαιο και αυτό είναι απαράδεικτο το να αναφέρεται σε αυτό το σώμα. Εμείς δεν το δεχόμεθα. Ο κύριος Κρίς Ντέβις. Πριν από τις μέρες ήμουνα στην ε, Γάζα. Ε, δεν είδα και πενταετή παιδάκια Ισραηλινά που αντιμετώπισαν τα όπλα των ε, Ναζί με τα χέρια πάνω από το κεφάλι τους. Σφιγγόταν η καρδιά μου αυτές τις φωτογραφίες. Και πώς επιτρέπουμε στο Ισραήλ πράγματα που δεν θα επιτρέπαμε σε άλλη χώρα. Αυτοί που τα λένε αυτά δεν εξηγούν γιατί αυτοί που υπέφεραν τόσο πολύ τον 20ο αιώνα κάνουν άλλους να υποφέρουν τόσο πολύ τον 21ο αιώνα. Διότι το Ισραήλ έκανε τη Γάζα κόλαση. Σύεται το έδαφος από τις εκρήξεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κατάβασης του πυρός. Και διάφορα κάρα, έχουμε κάρα στο δρόμο και F-16 στον ουρανό. Μηχανές του 20ου αιώνα που σκοτώνουν. Ρίχνουν βόμβες, 300 παιδιά πέθαναν, εκατοντάδες παιδιά έχουν διαλυθεί σε κομμάτια δεν είναι ανάλογη ανταπόκριση μιας πολιτισμένης δύναμης αυτή. Είναι κακό. Είναι κακό. Η δύναμη του κακού. Ναι, πρέπει να σταματήσουν οι πύραυλοι της Χαμάς. Το είπα αυτό στους εκπροσώπους της Χαμάς στη Γάζα, εγώ ίδιος. Αλλά μην κηρύττουμε, μην μιλάμε με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους για την ανάγκη πολέμης τρομοκρατίας. Διότι οι Παλαιστίνοι που βομβαρδίζονται θα μπορούσαν ε, να, κατο... να κατονομάσουν τον Όλμοντ και τον Λίβνε και τον Μπάρακ τρομοκράτες έχουμε κάποιες ευθύνες για τις δράσεις του Ισραήλ. Ποτέ κάτω παρελθόν, ποτέ, ποτέ, δεν μπορώ να σκεφτώ ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν στήριξε με κάποια δράση την κακή μεταχείριση, κακομεταχείριση των Παλαιστινίων από τους Ισραήλ, Ισραηλινούς. Δίνουμε το πράσινο φως στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και αυξάνουμε την αποτυχία αγνώντας τα μαθήματα της ιστορίας. Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη αν δεν μιλήσεις με τους εχθρού σου. Κι όμως αρνηθήκαμε να μιλήσουμε με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Παλαιστινιακού λαού. Και τώρα ολοκληρώνεται διαπραγματεύσει με το Ισραήλ για τη, διευρυμένη, για τη συμφωνία διευρυμένη συνεργασία. Δεν σχεδιάζουμε να καταδικάσουμε το Ισραήλ, αντιθέτω θέλουμε να τα ανταμείψουμε. Λοιπόν, εκείνοι που θέλουν δικαιοσύνη και για τις δύο πλευρές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ήρθε η ώρα ξανά να επανεξετάσουν το θέμα. Ο κύριο Ανέχτεν έχει για ένα λεπτό το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι σκανδαλώδες. Όλοι γνωρίζουν ότι μια στατιωτική λύση ποτέ δεν θα πετύχει στην Μέση Ανατολή. Η πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η συμφιλίωση σε αυτό το χώρο και πρέπει να τεθεί αμέσως τέρμα στις βιοπραγίες. Υποστηρίζω ε, τη δημιουργία ενός ανεξαρτήτου Παλαιστινιακού κράτους με τη δική του οικονομία, ε, με το δικό του πολιτικό σχέδιο. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρχουν δύο κράτη που θα σέβονται το ένα το άλλο. Το Ισραήλ σίγουρα έχει δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά νομίζω ότι πήγε πολύ μακριά με τις επιθέσεις του. Αυτές οι επιθέσεις είναι ανήθικες και η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Όταν η ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή θα πρέπει να αναζωογονηθεί αμέσως. Και ελπίζω ότι ο εκλογής πρόεδρο των ΗΠΑ ο Ομπάμα, θα δώσει τη δέωση προτεραιότητα στο θέμα και το εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το έργο και στην ε, μελλοντική του θέση. Ευχαριστώ. Χάμερσταϊν. Και εγώ παρευρέθηκα στη Γάζα όπου ζήσαμε μια ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία. Ζήσαμε και στην... Ε, πήγαμε, μεταβήκαμε και στην ε, Αίγυπτο. Λίγη η εποχή του Μπούς και βλέπουμε ότι οδηγεί, οδήγησε σε μία σφαγή. Θα πρέπει να προωθήσουμε μία νέα πολιτική στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την πολιτική του Ομπάμα, ο οποίος μας λέει ότι θα μιλήσει με το Ιράν και την Χαμάς. Πρόκειται για μια νέα πολιτική στη Μέση Ανατολή Θέλουμε να προωθήσουμε μια πολιτική συνεργασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει τις δικές μας αρχές και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Τα εκατοντάδες παιδιά στη Γάζα που μας κοιτούσαν στα μάτια με αυτές τις ματιές όλο ελπίδα. Αυτές τις εικόνες θα πρέπει να αποστείλουμε στο Ισραήλ. Αυτό σημαίνει επιτόπια δράση για να προωθήσουμε τους μετηριόφρονες γιατί ο Αμπτάλα, ο Μουμπάρακ και ε, άλλοι θεωρούνται προδότες. Ε, όταν εγώ μιλούσα με ορισμένους κατοίκους είδαμε είδαμε ότι υπήρχαν πολλές παράπλευρες απώλειες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την ειρηνευτική προσπάθεια, γιατί αυτή η παιδαγωγική της καταστροφής θα οδηγήσει στο μίσος. Και εσείς ξεπεράσετε κατά πολύ το χρόνο σας. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πόρτας ε, για ένα λεπτό. Μιλάμε για χίλιους θανάτους ε, μέχρι σήμερα. Πόσες ζωές θα στοιχήσει η εκλογή της Τζίπη Λίβνη και του Εχούντ Μπαράκ το Φεβρουάριο. Έχουν χαθεί πολλοί άμαχοι και εμείς όμως φέρουμε ευθύνη διότι το Συμβούλιο μίλησε για upgrading των σχέσεων με το Ισραήλ. Μιλάμε για συνέργεια εκ των προτέρων. Θα πρέπει να μιλήσουμε με την Χαμάς. Θα είχαμε κερδίσει πολύ περισσότερα αν είχαμε δεχτεί τις εκλογές και το αποτέλεσμα των εκλογών στην Παλαιστίνη. Δεν θα πρέπει να επικρατεί ο πιο δυνατός δεν πρέπει να χάνουμε ελπίδα. Θα πρέπει να γίνει κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτό εξαρτάται από το τέλος της κατοχής. Αυτή θα αυτό είναι το πραγματικό απτό αποτέλεσμα της ε, Realpolitik. Σύνοτι για ένα λεπτό. Αυτά που συμβαίνουν στην ε, Γάζα μας ε, λυπούν ιδιαίτερα, δηλαδή συνέχιση της καταστροφής από τη Δύση εγώ συμφωνώ 100% ότι οι Ισραηλοί έχουν το δικαίωμα να ζουν χωρίς την απειλή των επιθέσεων με ρουκέτες. Όμως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι ε, επιφορά δικαιοσύνης, ε, επιβολή δικαιοσύνης, αλλά είναι σφαγή. Το πιο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλα αυτά γίνονται από έναν ε, προτιμόμενο εμπορικό εταίρο για μας. Το 2007 είχαμε εμπορικέ συνταλλαγέ ε, πολλών δις ε, ευρώ και ως εκ τούτου ε, επειδή συμβάλλουμε τόσο πολύ στην οικονομία του Ισραήλ φέρουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη όταν τα χρήματα αυτά συμβάλλουν στο θάνατο των παιδιών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εμείς φέρουμε αίμα στα χέρια μας. Καλό λοιπόν όλους να επιβάλλουμε άμεσα εμπορικές κυρώσεις ε, εις βάρος του Ισραήλ και να παραμείνουν αυτές ε, μέχρι να επικρατήσει η κατάπαυση του πυρός. Αν δεν πάψουν οι δολοφονίες τότε και εμείς θα είμαστε συνεργοί στη σφαγή. Επόμενος ομιλητής, το κύριε Ζαΐφη για δύο λεπτά. Για άλλη μια φορά Δυστυχώς μίλησαν τα όπλα στη Μέση Ανατολή. Για άλλη μια φορά τα βασικά θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχουν τραυματιστεί χιλιάδες και σκοτωθεί εκατοντάδες. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται η ιστορία στις πύλες της Ευρώπης. Διαπιστώνουμε όμως ότι παρά αυτές τις πρωτοβουλίες η Ευρώπη δεν είναι αποτελεσματική για να επηρεάσει τα τεκτενόμενα. Αυτό είναι ακατανόητο γιατί για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινή γνώμης ε, η οποία αρνείται αυτή την ε, κατάσταση είμαστε αναποτελεσματικοί δεν είμαστε ηγετική δύναμη υπέρ της ειρήνης. Θα πρέπει να διαδραματίσουμε μείζωνα ρόλο και αυτό αφορά και την ε, ευρωμεσογειακή ζώνη και ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε άμεσα την ανακοχή και το άνοιγμα των σημείων διέλευσης καθώς και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού της Γάζας. Θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα, προωθώντας ε, μία ειρηνευτική δύναμη της Ευρώπης και της ευρύτερης Μεσογείου. Έτσι θα καταδείξουμε την πολιτική μας θέληση υπέρ μιας «παξ Europa που αναμένουν εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα όλοι οι λαοί της Μεσογείου. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή σε μια συνήθιστη κατάσταση. Με τη σύραξη αυτή μπαίνουμε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου. Δηλαδή στη σύραξη πολιτισμών, μεταξύ πολιτισμών. Υπάρχει πάντα μια κινητικότητα του αραβικού κόσμου. Τώρα όμως μιλάμε για κινητικότητα των μουσουλμάνων που ε, υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα. Η Ευρώπη φέρει ιστορική ευθύνη να ενισχύσει τον διάλογο των πολιτισμών. Βερονίκ Ντε Κάιζερ, δύο λεπτά και θα ήθελα να τηρήσετε και το χρόνο ομιλία σας, σας παρακαλώ. Πρόεδρε, Πολλές φορές έλαβα το λόγο εδώ στην Ολομέλεια έτσι ώστε να δράξουμε κάθε ευκαιρία για διάλογο γιατί έπρεπε να έχουμε προωθεί στο διάλογο με τη Χαμάς, η οποία στο κάτω-κάτω κέρδισε τις εκλογές. Δυστυχώς δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου δεν μπορώ παρά να εκφράσω τα συναισθήματά μου έναντι αυτής της φαγής, αυτής της προπαγάνδας, αυτού του αμήλικτου πολέμου. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα μίσους και αντισημιτισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα αίτια αυτής της κατάστασης η ζωή ενός Παλαιστίνιου ε, είναι αντίστοιχη με τη ζωή ενός Ισραηλινού και αυτό αφορά όχι μόνο τη ζωή του αλλά και το μέλλον του και την ελευθερία του. Δεύτερον, το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να τηρηθεί και αφορά την άμεση κατάπαυση του πυρός αλλά και όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό αφορά και τη σύμβαση της Γενέβης. Δυστυχώς όμως δεν επικρατεί το δίκαιο και οι λαοί βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας. Επίσης θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλα αυτά τα εγκλήματα, όποια και να είναι αυτά και από όπου και να προέρχονται. Ποτέ δεν θα υπάρξει ασφάλεια χωρίς ειρήνη, χωρίς, επίσης ειρήνη χωρίς ε, δικαιοσύνη και πιστεύω ότι γι' αυτό υπάρχει το δίκαιο και η δικαιοσύνη. Και πιστεύω ότι ένα δυναμικό, δυναμικό μια δυναμική πορεία υπέρ της ειρήνης θα πρέπει να οδηγήσει και σε εταιρικέ σχέσεις και στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί εξαίρεση, φέρει κρατική ευθύνη και θα πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο όπως και η Χαμάς. Δυστυχώς ο πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση ομοιρίας και εκατοντάδες παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους. Εμείς ως Ευρωπαίοι μπορέσαμε να φύγουμε από τη Γάζα, αλλά οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να φύγουν από τη Ράφα παρά μόνο αν είναι νεκροί ή τραυματίες, με φορεία δηλαδή. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτές τις βασικές αρχές λοιπόν. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, να τηρείτε το χρόνο που σας διατίθεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Θα ξεκινήσω απηχώντας αυτά που είπε ο κύριος Κονβεντίτ. Είναι η απελπισία που μας πνίγει σήμερα. Αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος, η τραγωδία. οι εικόνες των μαρτυρίων και των θανάτων ακατάπαυστα μας παρουσιάζονται στις οθόνες μας. Είναι κάτι αφόρητο και θέλω να πω ότι όλες οι εικόνες του πολέμου είναι τέτοιες, όλες οι συγκρούσεις και εκείνες που συζητούμε λιγότερα, για να μην πω που δεν αναφέρουμε Κονγκό, Νταρφούρ, Ζιμπάμπουε. Συγγνώμη. Και πριν από αυτό η Τσετσενία. Εκεί οι φρικαλαιότητε εξελίχθησαν και εξελίσσονται χωρίς να αναφέρονται από τα μέσα ενημέρωση και χωρί να τα συζητάνε οι πολιτικοί. ήδη εδώ επανειλημμένα είχα υπογραμμίσει εδώ την καταδίκη μου, μεταβλητή, την καταδίκη μεταβλητή γεωμετρία που εκφράζουν διάφοροι συνάδελφοι. Η κυρία Μαρκαντίνη το υπενθύμησε πολύ συχνά και εκείνη ότι δεν υπάρχουν λογιστικά στου θανάτου, δεν υπάρχει εράρχηση όσον αφορά τα μαρτύρια και το πώ υποφέρει κανεί. Κάθε νεκρό, παιδί, γυναίκα, παιδί και από τη μία και από την άλλη πλευρά είναι ένα θύμα παραπάνω. Τι να κάνουμε, ούτε στο σημερινή συζήτησή μα να μην είναι μια αντιπαράθεση άχρηστη και στήρα που συνήθω και ε, πώς θα ανταποκριθούμε στις ιστορικές μας ευθύνες. Μιλάω τελευταία ε, προ το τέλο τη συζήτηση, οπότε εξαντλήθηκαν τα επιχειρήματα σαν αφορά την κρίση του Ισραήλ, τη ελληνής απάντηση. Αλλά επουδενή όσον αφορά το δικαίωμα τη ασφαλεία του. Εν ονόματι. Μάλλον ε, θα, δεν θα μπορούσαμε να δεχόμαστε να βομβαρδίσει το Ισραήλ χωρί να αντιδρά. Χρειάζεται διαπραγμάτευση κατάπαυση του πυρός να υπάρχει ανθρωπιστική διέλευση, ανθρωπιστική βοήθεια να βρει διέλευση. Μέσω σειράγκων γίνεται αυτή τώρα. Πρέπει να εξεταστούν οι προοπτικές. Στην Τάμπα, στο Κάμπ Ντέιβιτ, στην Ανάπολη, σκιαγραφήθηκε κάπως η δίωδο για την λύση του προβλήματος. Χρειάζεται διαπραγμάτευση. Και οι δύο πλευρέ όμω θα πρέπει να παραιτηθούν. Τα μιλάω για παρέτηση, συμφωνώ με τον κύριο Σούλτ, που δεν είναι εδώ τώρα ε, όχι αν θα συνομιλήσει κανείς με τη Χαμάς ή όχι, αλλά πώς, υπό ποιες συνθήκες θα μιλήσει. Οι περισσότεροι συνάδελφοι μίλησαν 50 δευτερόλεπτα παραπάνω. Αφήστε με λοιπόν παρακαλώ να συνεχίσω. Το Μάιο του 1989 ο κύριος Σαραφάτ είπε ότι απαρνιέται ε, την προσέγγιση που μέχρι τότε μέσω της τρομοκρατίας και η συμφιλίωση χρειάζεται στην Παλαιστίνη. Και ρόλος μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί και άλλοι γείτονε, οι Άραβε, η Ορδανία και η Αίγυπτο να γίνουν εταίροι σε μια συμφωνία για βιώσιμη ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν ε, κάποιο ξεπερνάει το χρόνο του, ε, αυτό το κακό παράδειγμα που δίνει δεν πρέπει να το ακολουθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την ε, Κυριακή 11 Ιανουαρίου επισκεφτήκαμε το μεθοριακό σταθμό στη Ράφα, στην Γκάζα. Ε, που είναι αποκλεισμένοι. Δηλαδή οι πολίτες δεν έχουν καμία δυνατότητα να ξεφύγουν από την επίθεση των Ισραηλινών. Αν δεν έχει δει κανείς με δηλαδή τα μάτια δεν μπορεί να καταλάβει πόσο πολύ υποφέρουν οι άνθρωποι στη Γάζα και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να ξεβρεθεί μια λύση σε αυτή την σύγκρουση. Όλοι μας συγκινηθήκαμε αφάνταστα από τις ε, τεράστιες ταλαιπωρίες και τον πόνο των πολιτών των Παλαιστινίων. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ κατηγορηματικά να σταματήσουν πάρα αυτά οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών. Βεβαίως και να σταματήσουν και οι εκτοξεύσεις ρουκετών, ρουκετών από τη Χαμάς. Τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν πάρα αυτά έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάνει στον προορισμό της και να προσφέρεται στον άμαχο πληθυσμό. Στα σύνορα είδαμε ότι στεκόντουσαν ε, γιατροί εκεί σε αυτή την περιοχή για να μπουν στη Γάζα να προσφέρουν βοήθεια επειδή όμως τα σύνορα ήταν κλειστά δεν μπορούσαν να μπουν στη Γάζα. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ για άλλη μια φορά να ανοίξουν τα σύνορα έτσι ώστε πραγματικά η βοήθεια να φτάνει στον προορισμό της. Ε, Τσελέγγι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι παίρνουμε στα σοβαρά όλους αυτούς τους φόνους παιδιών και γυναικών. Ας μην είμαστε υποκριτές. Ποιε ευρωπαϊκές χώρες θα ήταν τόσο συγκρατημένε όσο το Ισραήλ εάν δεχόταν επίθεση επί σειρά ετών μέσω ρουκετών που απειλούν τη ζωή ε, πάνω από ένα εκατομμύρια πολιτών. Ναι. Λοιπόν, ε, ε, έχουμε τη Χαμάς που εξελέγει δημοκρατικά και μιλούσαν για απελευθέρωση. Δεν μιλούσαν όμω για απελευθέρωση τη γάζα, αλλά τη χάιφα και του Τελαβίβα από του Ισραηλινούς και ήθελαν την καταστροφή του Ισραήλ. Αν κάποιο ε, ψηφίζει εγκληματίε, πρέπει να μοιράζεται την τύχη των εγκληματιών. Κυρίω όταν οι εγκληματίε κρύβονται πίσω από τι πλάτε των αμάχων και εκτοξεύουν ρούκέτε από τζαμιά και σχολιά που τα μετατρέπουν σε πυρητή αποθήκες. Θυμάμαι το μοβαρδισμό της Δρέσδης που γκρεμίστηκαν τα πάντα από τους Βρετανικούς βομβαρδισμούς και δεκάδες χιλιάδες αμάχων ε, σκοτώθηκαν εξ αυτού. Κανείς δεν το επέκρινε αυτό, διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ταυτιστεί με τη μοίρα της Γερμανίας και ήξεραν ποιον ψήφισαν, όπως και οι Παλαιστίνοι που ψήφισαν τη Χαμάς. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη βοήθεια που πηγαίνει στη Γάζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Παλαιστίνοι στη Γάζα βοηθούμε αυτά τα χρήματα, ανοίγουν σύραγγε μέσω των οποίων περνάνε τα όπλα. Αυτό είναι δυσανάλογο. Γκούναρ Χόκμαρ για δύο λεπτά έχει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, υπάρχουν δύο σημαντικά ε, στοιχεία που καθορίζουν τη σημερινή συζήτηση. Πρώτον, ότι η συντριπτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, σε εμάς εδώ σήμερα, ζητάει την άμεση κατάπαυση του πυρός και δεύτερον όλοι υποστηρίζουν ότι το κράτος του Ισραήλ έχει δικαίωμα ύπαρξης έχει δικαίωμα να χαράξει ειρηνικά σύνορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την τραγωδία που βλέπουμε στη λωρίδα της Γάζας. Η ζωή που χάνεται είναι τραγωδία, ανεξάρτητα ε, σε ποιο ε, τμήμα, σε ποια πλευρά των συνόρων βρίσκεται. Και η τραγωδία δεν αμβλύνεται διότι οι μεν θέλουν να σκοτώσουν άμαχο πληθυσμό ή δεν ε, υποτίθεται μέλη της ε, Χαμάς. Είναι τραγωδία διότι με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται η ύπαρξη ειρηνικού κράτους του Ισραήλ. Είναι τραγωδία και για τη διεθνή κοινότητα, διότι με το λαθρεμπόριο όπλων κατέστη δυνατόν να υπάρξει αυτή η κατάσταση, η εκτόξευση των ρουκετών. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι η τραγωδία αυτή δεν προέκυψε από τη σύγκρουση ανάμεσα στους Εβραίους και τους Παλαιστινίους και εγώ ανθίσταμε στο να δαιμονοποιούμε ένα λαό όπως το έκανε ο κύριος Ντέιβις το να δαιμονοποιήσουμε πολίτες και λαό αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω ότι αρμόζει σε ένα κοινοβούλιο δεν πρόκειται για τη σύγκρουση ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Εβραίους αλλά πρόκειται για τη σύγκρουση ανάμεσα σε ακραίους και μετριοπαθείς πρέπει λοιπόν να πούμε την εκείνο που υποδαβλίζει το μίσος και σε εκείνους που το πράττουν αυτό πρέπει να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα επιτύχουν τίποτα. Αυτό πρέπει να το πει η Ευρώπη γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούν και οι μετριοπαθείς δυνάμεις να εργαστούν καλύτερα για την ειρήνη. Ο κύριος Μάρεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε εκείνους οι οποίοι αναφέρονται σε υποκρισία και δημαγωγία. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος ε, είναι μόνο άλλος ένας ε, πόλεμος ε, σε όλη αυτή τη σειρά των ασύμετρων επιθέσεων. Πριν λοιπόν από τον πόλεμο είχαμε επιθέσεις εις βάρος του Ισραήλ χωρίς να ενοχλείται κανείς. Τώρα όμως πολλοί στυλιτεύουν το Ισραήλ αυτό είναι μια απλούστευση γιατί κατ' ουσίαν έχουμε να κάνουμε ε, με μια κυβέρνηση, με ένα κράτος ε, που θα μπορεί η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Από την άλλη υποτίθεται υπάρχει ένα κράτος τρομοκρατών που δεν είναι απόλυτα γνωστό. Είναι συγκεχημένη κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με μια ασύμετρη κατάσταση κυρίως διότι από τη μία πλευρά έχουμε και άμαχο πληθυσμό που χρησιμοποιείται εν είδη ανθρώπινης ασπίδας. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Μόνο που όπως σας είπα έχουμε να κάνουμε και με ασυμμετρία όσον αφορά τις ε, λέξεις και τις πράξεις. Αν δεν υπάρξει διεθνής παρέμβαση, η σύγκρουση αυτή θα διαιωνίζεται στο διηνεκές. Ε, πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την άδικη επίθεση από πλευρά του Ισραήλ, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να γίνει όταν μία τρομοκρατική οργάνωση ε, από τη λωρίδα της Γάζας εξαπολύει ε, ρουκέτες εις ε, του Ισραήλ. Σίγουρα δεν είναι σωστή η αντίδραση του Ισραήλ γιατί αν το λέγαμε αυτό θα είχαμε να κάνουμε με ε, λέξεις που ε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο πρόεδρος, συνάδελφοι, τώρα πρέπει πραγματικά να σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο ε, που σας διατίθεται. Εγώ δεν σας διέκοψα, όμως ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Σβάτσενμπερκ, ε, διαθέτει περισσότερο χρόνο για μα από ό,τι θα μπορούσαμε να είχαμε ελπίσει. Θα είναι εδώ μέχρι τι 5 και 20, μου είπαν. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ να εστιάζετε την προσοχή σα σε αυτά που σα είπα. Το καλό παράδειγμα θα δώσει ο κ. Ε, Φιλίπ Μουριόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ειρηνευτική προσπάθεια, να καταπληθεί μια ειρηνευτική προσπάθεια. Στη Γάζα για πρώτη φορά το Ισραήλ φαίνεται να μην δέχεται ορισμένες βασικές αρχές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ειρηνευτική δύναμη θα μπορέσει να εγκατασταθεί εκεί όταν επιληθεί η σύραξη αυτή. Γνωρίζω ότι αυτή αποστολή σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αμεροληψία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση για να αναλάβει δράση και στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Ένωσης θα μπορέσει να δράσει γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Αμερικανοί είναι υπέρ των Ισραηλινών και οι Άραβες υπέρ των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες διχοτομήσεις. Δεν θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά. Ευχαριστούμε που τηρήσατε τον χρόνο. Επόμενος ομιλητής ο κ. Ζαλέσκη για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η, η κατοχή τελικά δίνει καρπούς, αναποτελεσματικότητα των αρχών, οργή και τη συνέπεια αμάς, το αποτέλεσμα αμάς όπως θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε, σοβαρός παράγων. Απαράδεκτο είναι ότι οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι και οι Χαμάς αρνούνται το Ισραήλ, καθώς και ότι χρησιμοποιούν σαν ασπίδες τα παιδιά. Δεν επιτρέπεται συνεχής απειλή να στρέφεται κατά των Ισραηλινών παιδιών φαύλος κύκλος είναι επιθετικότητας. Οι ζαϊνές αρχές μπορούν να πάρουν τα μαθήματά τους από την εξαετία που πέρασε στην περιοχή και να χωρίσουν ε, την περιοχή σε δύο χώρες. Σαν επιχείρηση με νηστέρι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να δεχτούν να γείτονα επεκτοξεύει πυράβλους. Αλλά οι διεθνεί κοινότητε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσω μπορέσουν να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση. Είναι μια, η λύση που προτείνεται αποδεκτή σήμερα από το Ισραήλ. Υπάρχει άλλη λύση όμως. Αν υπάρχει προτείνεται το. Να περιμένουμε να πεθάνουν όλα τα μέλη της ε, Χαμάς ή να τους βομβαρδίσουμε να σκοτωθούν όλοι. Αυτό δεν στέκει. Χρειάζεται περισσότερο θάρρος από πλευράς Ισραήλ. Αν οι δυτικές δυνάμεις δεν δημιούργησαν δύο κράτη το 1948 θα πρέπει να το κάνουν τώρα.

στόχος είναι να καταστραφεί η Χαμάς ε, ο αποδεκατισμός ε, της ε, Χαμάς όμως οδηγεί στο να σκοτώνται και Ισραηλινοί. Στο επίπεδο και στην πλευρά των Παλαιστινίων σκοτώνονται άμαχοι πολίτες. Αυτοί δεν είναι μέλη της Χαμάς. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να επιτευχθεί και χειρία αν το, η μία οντότητα δεν αναγνωρίζει την άλλη θα πρέπει ε, το υποκείμενο της επίθεσης να καταστεί αντικείμενο και τα νάπαλη και αυτά για να καταστεί δυνατή η τήρηση και ο σεβασμός της ειρήνης. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τη Χαμάς και να ξεκινήσουμε το διάλογο. Και τα Νάπαλη, η Χαμάς πρέπει να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένας, καμία λύση. Ε, όλοι οι πόλεμοι είναι καταδικαστέοι. Ε, πρέπει να δώσουμε το πάνω χέρι στην ε, πολιτική. Ο κύριος Όλμερτ, ο Ισραηλινός, προσπαθεί να βελτιώσει το κύρος του, ε, αλλά δεν επιτρέπει την εκεχηρία. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο, Η κυρία Ιμπάσκοβα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα ε, να σας ε, συγχαρώ θερμά για τα αποτελέσματα τα οποία επιτύχατε με την αποστολή στο Ισραήλ. Με τη δική σας ε, τη βοήθεια κατέστη δυνατόν ε, να πιστεί το Ισραήλ να ανοίγει για τρεις ώρες ε, τα σημεία διέλευσης. Νομίζω οι Ισραηλοί για πρώτη φορά λαμβάνουν ε, σοβαρά υπόψη τους ε, τους Ευρωπαίους ε, και λαμβάνουν υπόψη τους και τους Τσέχους ε, οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν μια λύση με τη Χαμάς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τεταμένη και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει μια, ένα ισόρροπο ψήφισμα. Και νομίζω ότι ένα τέτοιου είδους ε, ψήφισμα πράγματι το έχουμε επιτύχει. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ή μάλλον η Χαμάς πρέπει να αναγνωρίσει το Ισραήλ ως κράτος. Πρέπει να πάυσει να εκτοξεύει ρουκέτες ε, ενάντια σε αυτό το κράτος και η κατάπαυση του πυρός πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινοί Πρέπει ε, λοιπόν να αποδείξουν ε, κάτω από ποιες συνθήκες είναι πρόθυμοι να σταματήσουν τις στρατιωτικές τους επιθέσεις. Νομίζω η Αίγυπτος ε, καλύτερα να εμπειρωματεί σημαντικό ρόλο, παραδείγματος χάρη να αναχαιτήσει το λαθρεμπόριο όπλων. Το Συμβούλιο Πώς ακριβώς συμμετέχει το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις ε, με τους Αιγύπτιους, πώς αντιμετωπίζονται θέματα του ε, τεχνικού ελέγχου. Εμείς οι Ευρωπαίοι τι μπορούμε να ζητήσουμε από τους Αιγύπτιους. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Αυτά όλα είναι θέματα που είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενη ομιλήτρια, επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Ρούτσεκ, Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να κάνω έκκληση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση και προς τα δύο μέρη της ε, σύραξης. Έχουμε την, ε, το ψήφισμα 1860 των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θα πρέπει να τηρήσουμε. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε μία μακροχρόνια εκεχηρία για να ανοίξει και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος Καμία στρατιωτική λύση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από πολιτικές διαπραγματεύσεις σε συνεργασία και με τον Αραβικό Σύνδεσμο και της ΕΠΑ που διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή η μακροχρόνια διένεξη θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση που να εμπεριέχει δύο κράτη έτσι ώστε να μπορέσουν οι δύο λαοί να ζήσουν από κοινού ειρηνικά ε, σεβόμενοι αμοιβαία τα σύνορά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κασουλίδης για δύο λεπτά. We are yet another... Συζητάμε άλλη μια ανθρωπιστική τραγωδία στη γειτονιά μας, δίπλα στη χώρα μου, όπου οι δύο τέροι μας στην ε, Μεσόγειο έχουν αναμειχθεί. Δυστυχώς οι Παλαιστίνοι δεν έχουν δεχτεί ακόμα ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας και οι πύραυλοι Κασάμ ποτέ δεν θα τους απελευθερώσουν από την κατοχή. Το Ισραήλ δεν καταλαβαίνει απ' την άλλη ότι τέτοια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση δημιουργεί ενδεχομένως νέους υποψηφίους για επιθέσεις αυτοκτονίας και νέες εκτοξεύσεις Κασάμ. Τι γίνεται με τους αθώους πολίτες, τους άμαχους, γυναίκες, παιδιά. Κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς. Κανείς δεν νοιάζεται για τα παιδιά που σκοτώνονται, ακροτηριάζονται, καίγονται, τραυματίζονται εκατοντάδες. Τα παιδιά του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Εμείς από την άνεση του καναπέ και της τηλεόρασης αισθανόμαστε ναυτία βλέποντας όλα αυτά. Σκεφτείτε αυτοί που είναι εκεί, πώς αισθάνονται. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να αρχίσουμε να κατηγορούμε. Αυτό δεν βοηθάει τους άμαχους. Να περνάμε ψηφίσματα, ούτε αυτό βοηθάει τους άμαχους. Από τα λόγια πώς περνάμε στις πράξεις. Τώρα ήρθε η ώρα να διαπραγματευτούμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να διαμορφωθεί μια διεθνής δύναμη, όπως πρότειναν και άλλοι συνάδελφοι, που θα πάει στη Γάζα. Με μεγάλη νομική συνιστόσα που θα ανδρώνεται από αραβικές χώρες. Και θα συμμετέχει και η Παλαιστινιακή Αρχή και η αστυνομική της δύναμη. Και εντολή των Ηνωμένων Εθνών θα δοθεί σε αυτή τη δύναμη. Και η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Δύναμη θα πάει για να θέσει τέρμα στην εκτόξευση των ρουκετών στο λαθρεμπόριο όπλων και να ανοίξουν τα σημεία διελεύσεως. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η μοίρα των αμάχων πλέον να βρίσκεται στα χέρια των δύο αντιθέτων πλευρών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιέζα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, μεγάλο αντιφασή Ιταλό, ο Πιέρο Γκομπέτη, είχε πει ότι όταν η αλήθεια είναι με τη μία πλευρά, μια σολομόντια λύση ε, είναι τελείω. δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Το ίδιο και για τη Γάζα αυτέ τι μέρε. Ελπίζω αυτό το κοινοβούλιο να μπορεί να πει αρκετά λόγια για να μπορεί να σταματήσει το Ισραήλ. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα καλυφθεί από ντροπή έναντι τη ιστορία, έναντι των Παλαιστινίων, έναντι τη ευρωπαϊκή δημόσια κοινή γνώμη και τη αραβική. Το Ισραήλ βομβαρδίζει και αποδεκατίζει ένα γκέτο. Εκείν, τα παιδιά εκείνων που καταστρέφονται γίνονται εκείνοι καταστροφή. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Έχει δικαίωμα στην ασφάλεια το Ισραήλ. Μπορεί να δει κανείς όποιος θέλει ότι κανένας δεν μπορεί να απειλήσει το Ισραήλ και την ύπαρξή του. Το βλέπουμε από την ισορροπία των δυνάμεων στο στρατό, στην πεδίο της μάχης. Το βλέπουμε από τον απολογισμό νεκρών και τραυματιών. την υποστήριξη που δίνει η Δύση στο Ισραήλ. Λοιπόν, δεν έχει άλλο σκοπό αυτή η επίθεση παρά να εμποδίσει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι σκοτώνεται η ειρήνη. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε το Ισραήλ. Στέφανο Τσάπαλα, ο κύριος Σαπαλά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα, τον Υπουργό Εξωτερικών, διότι είναι ακόμα μαζί μας. Κάτι στο οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι. Η συνάδελφος Μουσκαρντίνη έχει δίκιο. Όποιος δεν γνωρίζει ε, τη χωροταξική κατάσταση δεν μπορεί να ε, αρθρώσει σαφή και ακριβή λόγο. Δηλαδή θα ήταν σκοπιμότερο να μεταβεί εκεί. Όχι βεβαίως για, καθαρά, για λόγους ε, τουρισμού. Όπως ξέρετε είχαμε παρευρεθεί εκεί για τις εκλογές του Αμπού Μάζεν στο παρελθόν και ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Ε, αυτή η πείρα μας είναι δεκαετής τουλάχιστον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το θεωρούμε σαν ένα γεγονός που αφορά δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Εγώ έχω μεταβεί στο Ισραήλ πολλές φορές, γνωρίζω αρκετά καλά την κατάσταση και εδώ μπορούμε να πούμε ότι στο πρόβλημα αφορά, το πρόβλημα αφορά του τρομοκράτες, το κράτος του Ισραήλ και ε, ο λαός της Παλαιστίνης είναι το ενδιάμεσο θύμα. Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό. Εγώ αναφέρθηκα σε όλα τα θύματα και δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, μεγάλη, δηλαδή δεν μπορούμε να ταυτίσουμε την ε, λωρίδα της Γάζας με την Δυτική Όχθη. Είδα και ένα φιλμ επί του θέματος και γνωρίζω πώς έχει κατάσταση. Και σήμερα έχει αποδυναμωθεί ο Αμπού Μάζεν, ο οποίος είναι πιο αποδυναμωμένος παρά ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που χάνουν είμαστε όλοι εμεί. Κυρία Κοπά, ένα λεπτό. Η γνώμη σε όλη την Ευρώπη ζητά ένα πράγμα από την Ένωση. Βάλτε τέλο στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Πρέπει να καταδικάσουμε την τυφλή βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά και να είμαστε συνεπεί αναγνωρίζοντα ότι το Ισραήλ απαντά με κρατική τρομοκρατία μαζική κλίμακα. Η ασύμετρη ανταπόδοση, η καταπάτηση κάθε έννοια διεθνού και ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρου του Ισραήλ δεν μπορεί να γίνει ανεκτή είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται βόμβες λευκού φωσφόρου και άλλα πειραματικά όπλα κατά μάχων και είναι απάνθρωπο να στοχοποιούνται αθώες γυναίκες και παιδιά. αν αυτό συνέβαινε στην αφρική ή σε άλλο μέρος του κόσμου η αντίδρασή μας θα ήταν άμεση και η απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας δεσμευτική. στην περίπτωση του ισραήλ όμως περιοριζόμαστε σε δηλώσεις και ατελέσφορες συζητήσεις πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πολιτικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης ώστε να πιστεί το ισραήλ να σταματήσει την παράλογη βία εναντίον του παλαιστινιακού λαού αλλά και την απαγόρευση πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας. δεν μπορούμε να είμαστε αμέτωχοι θεατές γιατί έτσι γινόμαστε συνυπεύθυνοι στη σφαγή. η μόνη λύση είναι η άμεση πάυση πυρός και το άνοιγμα ανθρωπιστικών διόδων προς τη γάζα αλλά και η έναρξη διαλόγου με όλες τις πλευρές. Ε, κύριος ε, Στίβενσον για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, τα τραγικά γεγονότα στη Γάζα τις δύο τελευταίες εβδομάδες ε, οδήγησαν στο να καταδικάσουμε διεθνώς το Ισραήλ. Σήμερα όλοι οι συνάδελφοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους απέναντι στο εβραϊκό κράτος. Όμως για ένα κράτος στη Μέση Ανατολή αυτό ακριβώς ήθελαν. Δηλαδή το Ιράν έδωσε τους πυράβλους και εξελιγμένα όπλα στη Χαμάς εδώ και χρόνια. Έχουν προσφέρει την εκπαίδευση χρήματα ε, στη Χαμάς με στόχο να προκαλέσουν το Ισραήλ να ξεκινήσει αυτό το πόλεμο και βλέπουμε αυτές τις εικόνες στις τηλεοράσεις, τα εμόφυρτα παιδιά και σε εφημερίδες και αυτό αν θέλετε είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσιλητιστούν οι φανατικοί μουσουλμάνοι έτσι ώστε να υπάρχει μια παγκόσμια μουσουλμανική κίνηση ενωμένη κατά της Δύσης. Το φασιστικό καθεστώς του Ιράν είναι ο βασικός χρηματοδότης ε, της κατάστασης ε, στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς ήθελε το Ιράν ε, αποσπά την προσοχή από την οικονομική κρίση του Ιράν λόγω και της κατάρρευσης της ε, τιμής του πετρελαίου και επίσης και από τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα για να έχει πυρηνικά όπλα. Ε, στόχος είναι του Ιράν να γίνει κυρίαρχη δύναμη, θέλουν να ενώσουν τον μουσουλμανικό κόσμο κάτω από το δικό τους το όραμα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, μιας μουσουλμανικής αδελφότητας όπου ε, δεν θα υπάρχει δικαίωμα λόγου και δυστυχώς ε, η Δύση δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική επίθεση. Η Δύση δυστυχώς ε, το ανάντιο έκανε, προσπάθησε να καθησυχάσει το Ιράν και δεν στήριξε αρκετά την αντιπολίτευση ε, γιατί ε, δυστυχώς ε, τους έθεσε και στην λίστα των τρομοκρατών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ο κύριος Χάουιτ. Κοιτάξτε, σήμερα το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει το ψήφισμα του ΟΗΕ 1860 και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το ψήφισμα αμελητή. Και σαν ένα από του ευρωβουλευτέ που έχει πάει στη Γάζα κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, μια κατάπαυση του πυρό και απόσυση δεν αρκεί. Ναι βεβαίω θέλουμε να σταματήσουν οι εκτοξεύσει των ρουκετών και να σταματήσουν τι κινήσει του τρομοκράτε, αλλά πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρό και τερματισμό του αποκλεισμού του, ώστε ο λαό τη Γάζα να ζει στη ζωή του. Είναι ένα θέμα σεβασμού του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, η Human Rights Watch και η ε, Islamic Relief μου είπαν ότι η τριετή διακοπή είναι άκρως ανεπαρκής για να διανεμηθεί βοήθεια και είναι θέμα αναλογικότητα. Η Save the Children λέει ότι 139 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη των ε, εχθροπραξιών και 1.271 παιδιά τραυματίστηκαν. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό άμυνα. Και τέλος, Πρόεδρε, καλωσορίζω τη σημερινή δήλωση ότι ο κ. Συμπριάνο Ζαλ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σταματά, παγώνει τις συζητήσεις για αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Για αυτούς τους λόγους και αυτό έπρεπε να κάνουν. Για δύο λεπτά, κύριος Γκάλερ. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ε, κατάπαυση του πυρός σε διαρκείες και στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι αυτού συμφωνούν ε, όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ε, διεθνή κοινότητα πρέπει να ασχοληθούμε με τη μοίρα ε, των λαών, των πολιτών της Γάζας. Να μην το αφήσουμε τη μοίρα τους στις δύο πλευρές. Η Χαμάς ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μακροπρόθεσμα το Ισραήλ θα αντιδρούσε στις ρουκέτες και όχι μόνο λόγω προεκλογικής εκστρατείας. Πέρυσι οι σφιγμετρήσεις επιχειρήσεις έδειξαν ότι πέφτει η Χαμάς και ανεβαίνει η Φατάχ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η Χαμάς αποφάσισε με ε, τα θύματα αυτά να αυξήσει και πάλι την επιρροή της. Κοινικό αυτό, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ ε, έχει κατά νου μόνο τα συμφέροντα των δικών του των ε, πολιτών. Η κριτική που ασκείται σε διεθνές επίπεδο αφορά κυρίως την έκταση της επιχείρησης και το γεγονός ότι σκοτώνουν τόσοι πολλοί άμαχοι. Γι' αυτό λοιπόν ως Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο άλλη μία κατάπαυση πυρός και τη χρηματοδότηση της ε, υποδομής. Ήδη βλέπω ότι θα υπάρχει μία διορθωτική επιστολή της Επιτρόπου που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και δεν αρκεί ε, να αναθέσουμε στους Αιγύπτιους ε, για να ελέγχουν αυτοί κατά πόσον θα υπάρχει λαθρεμπόριο όπλων ή όχι. Εγώ ε, απαιτώ οι τετραμερείς όπου θα συμμετέχουν και περισσότερες αραβικές δυνάμεις όλοι από κοινού στη Γάζα να επέμβουν με στρατιωτικές δυνάμεις έτσι ώστε να υπάρχει διαρκή ειρήνη και αυτό προς όφελος των πολιτών της Γάζα, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Και παράλληλα η ειρηνευτική διεργασία πρέπει να συνεχιστεί ταχύτατα γιατί αλλιώ φοβάμαι ότι όλο και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα θα έχουμε γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στη Γάζα και αυτό δεν αξίζει ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Παλαιστίνιους. Ευχαριστούμε που κρατήσατε τον χρόνο σας. Ο κύριος ε, Μαρτίνες Μαρτίνες. Μαρτίνες έχει το Εμείς οι Ισπανοί ζούμε αυτήν την κατάσταση της ε, Γάζας ε, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μας. Πιστεύουμε ε, βλέποντας αυτές τις εικόνες των αιμόφυρτων, των νεκρών, των βομβαρδισμών ότι στην Κερνίκα του Πικάσο αποδίδεται πολύ σωστά αυτή η φρίκη και ο αποτροπιασμός. Ε, εκφράζουμε την τροπή μας διότι δεν καταφέραμε ως διεθνής κοινότητα να προλάβουμε την κατάσταση ή να την αντιμετωπίσουμε. Ε, νιώθουμε ντροπή και αποτροπιασμό γιατί γνωρίζουμε επακριβώς τι συμβαίνει και δεν δρούμε με την κατάλληλη πιστικότητα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εγκληματική αυτή κατάσταση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε το ψήφισμα που ήρθε αργά του Συμβουλίου Ασφαλείας και να λάβουμε υπόψη και τις διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ. Βεβαίως και η Χαμάς ε, είναι υπεύθυνη γιατί δεν άκουσε κανέναν, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Χαμάς. Παν mm. Όρντεν για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την κάθε, τη συμπόνια μου προς όλους αθώους και στο Ισραήλ και τη Γάζα που υποφέρουν στους τελευταίους μήνες και μέρες. Ο, αλλά υπάρχουν όμως οι διάφορε ανησυχίε. Βέβαια, αλλά καταλαβαίνουν ποια είναι η πραγματική φύση τη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Στη Γάζα η Χαμά δημιούργησε μια επικράτεια τρομοκρατική. Δεν ανέχεται καμία αντιπαλότητα απόψη τη. Δολοφόνησε του Παλαιστινίου που ήταν αντίθετοι. Χώρισε την Παλαιστινιακή Αρχή σε κομμάτια και ε, επιτίθεται κατά των Ισραηλινών πολιτών, αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, αρνείται να δεχτεί τις πρώτερες συμφωνίες ειρήνης. Ο Χάνα Νασράουιτ είχε πει πριν τρία χρόνια όταν εγώ έλεγχα τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Χάναν. Ε, οι δυνάμεις του σκότους επέβαλαν τον νόμο. Αυτό, αυτό έβλεπε. Είχε πολύ δίκιο. Α μην εκπλησόμεθα ότι ένα βουλευτή τη Χαμά υπερηφανευόταν όταν λέγει ότι ο θάνατο ήταν μια βιομηχανία για τον Παλαιστινιακό λαό αναφερόταν στη χρήση των επιθέσεων αυτοκτονίας και την χρήση ανθρωπίνων ασπίδων αμάχων για την προστασία στρατιωτικών στόχων. Αυτό είναι παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να χρησιμοποιεί κανείς αμάχους του το τρόπος. Αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο φρικτό εχθρό, τι να κάνει το Ισραήλ όταν απειλούνται οι πολίτες του, και δέχονται τρομοκρατικέ επιθέσει. Η διεθνή κοινότη δεν το σημείωσε επαρκώ αυτό. Όταν το Ισραήλ έδρασε χωρί βία, επιβάλλοντα αποκλεισμό, κόβοντα το ηλεκτρικό ρεύμα, καταδικάστηκε. Τώρα που κινήθηκε στρατιωτικά, ανταποκρινόμενο στι προκλήσει του Ισραήλ, δέχεται την παγκόσμια κατακραυγή. Ποια είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Ότι ο Παλαιστινιακό λαό επί σειρά ετών καταπιέστηκε από εκείνους που ελέγχουν την Παλαιστινιακή Αρχή από τη διεθνή κοινότητα που έχει ανεχθεί τη διαφθορά και τι ακρεφνεί θέσει και από τον αραβικό κόσμο που επί σειρά δεκαετιών δεν έκανε κάτι πρακτικό για να βελτιώσει τη ζωή του και την προοπτική του. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Marshall για τη Μέση Ανατολή. Οι Παλαιστίνοι δεν χρειάζονται απλώ ειρηνευτέ, αλλά σωστή διοίκηση, χωρί διαφθορά. Και αυτή η διοίκηση θα πρέπει να ελέγχεται από διεθνή φορέα αλλά πρέπει να αποκόψουμε τους δημοκρατές, όπλα, χρήματα και πολιτική ανοχή. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντερόσα έχει το λόγο για ένα λεπτό μετά τον κ. Βανόρντεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κ. Βανόρντεν ε, για τη Χαμάς. Είναι όμως ε, γεγονός ε, ότι τίποτα από αυτά που είπε δεν ε, δικαιολογεί τον βομβαρδισμό αμάχων από πλευρά του Ισραήλ. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Είτε έρχονται από τη Χαμάς είτε από το Ισραήλ. Ελπίζω ότι το ψήφισμα μετά τη συζήτηση θα υπερψηφιστεί σε μεγάλο βαθμό από τους περισσότερους και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να σταματήσουν οι δολοφονίες στη Γάζα. Γιατί η περιοχή αυτή έχει γίνει η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει γίνει μάλιστα και σφαγείο η Γάζα. Η Γάζα χρησιμοποιείται η τρομοκρατία κατά της ε, τρομοκρατίας, δολοφονούνται άνθρωποι και παιδιά και έτσι δολοφονείται και η ελπίδα να υπάρξουν στο τέλος δύο κράτη. Δεν μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ όσο το Ισραήλ δεν έχει επικοδομητικές σχέσεις με τις όμορες χώρες και με τους ερετούς Παλαιστινίους συμπεριλαμβανομένης και της Χαμάς. Η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα θα υπάρξει και κλιμάκωση κλιμάκωση των δικών μας των αντιδράσεων. Η κυρία Γκάλ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία, κυρία Επίτροπε. Είναι κοινικός ο τρόπος συζήτησης της ε, κρίσης ε, στη ε, Γάζα. Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως ανθρώπινη ασπίδα, ιδιαίτερα παιδιά και είναι ιδιαίτερα κοινικό αυτό. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για μη αναλογικά ε, μέτρα τη στιγμή που σκοτώνονται πολλοί άμαχοι. Νομίζω ότι αυτό αφορά και την διεθνή διπλωματία, διότι δημιουργεί αυταπάτες. Μιλάμε επίσης και για ανθρωπιστική βοήθεια προς τα θύματα. Εγώ υψώνω τη φωνή μου υπέρ των παιδιών, γιατί δεν, ε, δεν μπορεί να εξηγηθεί και να δικαιολογηθεί ποτέ ε, ο σκοτωμός αμάχων και ιδιαίτερα παιδιών για οποιοδήποτε σκοπό και αυτό αφορά παιδιά οπουδήποτε και αν ζουν, σε όποια πλευρά των συνόρων και αν ζουν. Η προστασία των πολιτών αποτελεί αξία καθεαυτή και η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να προωθηθεί για να επιτευχθεί και μία μακροχρόνια και χειρία για να οδηγήσει στην, σε μία μακροχρόνια ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκάλ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ. Η Χαμάς προωθεί την τρομοκρατία και τα αντίπεινα. Φαίνεται λοιπόν ότι πολλοί ε, προωθούν παιδιά μάρτυρες και έτσι με αυτή τη δημοσιότητα προωθούν τη δική τους υπόθεση. Αυτό είναι ικτρό. Εγώ ποτέ δεν υποστήριξα την τρομοκρατία το Ισραήλ έχει το δικαίωμα ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή, αλλά βεβαίως ε, εκφράζουμε την τροπή μας για το τι συμβαίνει επί του παρόντος στη Γάζα, διότι ε, ε, δεν είναι αναλογική η απάντηση του Ισραήλ και ο θάνατος μικρών παιδιών είναι ντροπιαστικός. Πιστεύω ότι οι συμβουλές του Δαλάη Λάμα ήταν ε, οι καλύτεροι. Δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις που θα πρέπει να προωθηθούν και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την κλίμακα των γεγονότων. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανθρωπιστικές ανάγκες ε, της περιοχής και το γνωρίζουμε αυτό στη κοινή συνεδρίαση της ΑΦΕΤ και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα θέλαμε να προωθηθεί ένα εκτενές πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας για να κινηθούμε προς τα εκεί και να βοηθήσουμε τα θύματα με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σφάρτσεμπεργκ. Εάν βιάζεστε και θέλετε να παρέμβετε τώρα, μπορείτε να το κάνετε και μετά θα έχουμε τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Μετά θα έχουμε τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Θα πρέπει να απαντηθούν πολλά και διάφορα ζητήματα ύψης της σημασίας. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή ήταν το εξής. Κατά πόσο θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη Χαμάς. Δεν νομίζω ότι ήρθε ο καιρός γι' αυτό. Η Χαμάς ε, τους τελευταίους μήνες ε, συμπεριφέρθηκε έτσι ώστε να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Τη στιγμή που είναι αυτή η συμπεριφορά της δεν μπορούμε να έρθουμε επίσημα σε επαφή με αυτήν ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, μακροχρόνια πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις αλλάζουν συμπεριφορά και στο τέλος μπορούμε να τις αποδεχτούμε ως ε, διεθνής κοινότητα. Το είδα στην Αφρική, στην Ιρλανδία και σε πολλά μέρη. Αυτό συμβαίνει. Αλλά καταρχήν θα πρέπει να μην δρουν πλέον ως τρομοκρατική οργάνωση. Μετά θα είμαι έτοιμος να έρθω σε επαφή με τη Χαμάς, αλλά όχι πριν δεν μπορούν να δρουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απαρνηθεί τις αρχές της. Δεν μπορούμε να δεχτούμε έμεσες επαφές ερχόμαστε σε επαφή με πολιτικούς της ευρύτερης περιφέρειας, αλλά δεν ήρθε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε επαφή με την Χαμάς άμεσα. Θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι ως προς αυτό. θα πρέπει να επενέσουμε την Αίγυπτο για το σημαντικό της ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες, γιατί εργάζεται πολύ σκληρά για την κατάπαυση του πυρός και για μία ανακοχή ενδεχομένω. Και βέβαια για την ειρήνευση στην περιοχή. Γνωρίζω ότι το ζήτημα είναι πολύ δυσχερές. Είμαστε σε επαφή με τους Αιγύπτιους. Γνωρίζουμε την επίπονη εργασία τους και θα θέλαμε να τους συγχαρούμε. πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ευρύτερη περιφέρεια. Αυτοί που βρίσκονται επιτόπου θα πρέπει να μας πούνε ποιες είναι οι ανάγκες τους. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς τι θα τους δώσουμε. Θα πρέπει να μας το ζητήσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά κράτη της τόνισαν την ετοιμότητά τους να παρέμβουν, δηλαδή να αποστείλουν συμβούλους, να προετοιμάσουν τα κατάλληλα μέσα, αλλά βεβαίως με την συνένεση των ενδιαφερομένων εκεί, στην ευρύτερη περιοχή. θα είχα να προβώ και σε μία υπόδειξη, δηλαδή να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα Marshall για την ε, περιοχή αυτή. Πολύ καλή είναι αυτή η ιδέα, πράγματι. Χρειάζεται μία ανοικοδόμηση ε, αυτή η περιοχή και αυτό το σχέδιο Marshall που βοήθησε την Ευρώπη μετά από τον πόλεμο θα μπορούσε να βοηθήσει και τη Μέση Ανατολή. Η κυρία Φερέρο Βάλντνερ μίλησε για τις επιμέρους αποστολές. Επιτύχαμε πολλά και θα ήθελα να επενέσω την κυρία Φερέρο Βάλντνερ διότι ήταν επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας και προσπαθήσαμε να επιδώσουμε και ανθρωπιστική βοήθεια. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και είναι δυσχερείς. και τις ανάγκες αυτές τις είχαμε διαπιστώσει και στην Εγγύς Ανατολή. Εκεί είχαμε έρθει σε επαφή με τους εταίρους μας και είδαμε ότι το σχέδιο ήταν επιτυχές. Μιλήσαμε για το upgrading, για τη βελτίωση των σχέσεών μας με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια απόφαση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο πέρυσι. Και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο εάν οι Υπουργοί αλλάξουν αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί να αλλάξει από εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιερουσαλήμ. Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση, η αναβάθμιση των σχέσεων μας με το Ισραήλ και αν θα οργανωθεί μια διάσκεψη κορυφή στο εγγύς μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίγοντα ζητήματα προς αντιμετώπιση και θα ήθελα να πω ότι η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Υπουργών και δεν μπορεί να αναιρεθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε το Ισραήλ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολύ λίγα. Το Ισραήλ δρά κατά τον τρόπο που δρά και επειδή είμαι φίλος του Ισραήλ αναφέρω ειλικρινά ότι δεν είμαι και τόσο ευτυχής με το πώς δρούν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ λίγες δυνατότητες πέρα από τη δύναμη του λόγου. Σας μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια και μιλώ έτσι και στους εταίρους μας. Τη λύση θα πρέπει να την εξεύρουν οι εταίροι στην Εγγύης Ανατολή, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο μετά την κατάπαυση του πυρός. θα πρέπει να κλείσουν και τις σύραγγες όπου περνάνε όπλα στη λωρίδα της Γάζας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε με την διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων αλλά δεν έχουμε τη δύναμη και τα μέσα να σταματήσουμε τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να αποστείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή αυτή. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και οι δύο πλευρές εξαρτώνται από άλλες δυνάμεις το Ισραήλ έχει και άλλους συμμάχους εκτός Ευρώπης. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες, αλλά τίποτα άλλο. Και έτσι ε, μπορούμε να επιτύχουμε μερικά πράγματα, αλλά ας μην υπερβάλλουμε ως προς τις δυνατότητές μας. Ωραία, περνάμε στις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Ο κύριος Καρίμ έχει το λόγο για ένα λεπτό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 Πράγματι αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Αν αυτό ισχύει τότε ε, θα πρέπει να ισχύει και η αρχή της αναλογικότητας. Το γεγονός ότι το Ισραήλ τα αγνοεί αυτά είναι σαφές ε, και το να το γνώμη όμως εμείς αυτό είναι λάθος. Η χρήση λευκού φωσφόρου εις βάρος ε, των αμάχων αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε που την αντιδράστηκε ο μένοντας πολιτιών δεν επιρρίξει. Και αυτό είναι άδικο. Ο χρόνος, ο χρονισμός ήταν πολύ καλά υπολογισμένος από πλευρά Ισραήλ. Φτάνει 20 Ιανουαρίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο απόλυτη κατά του Ισραήλ. Θα δεχθούμε λοιπόν αυτό να ξαναγίνει. Θα υπάρξει συνεργασία μαζί μας ε, για να λυθεί το πρόβλημα. Οι Παλαιστίνοι ρωτούν πώς είναι δυνατόν η χώρα σας να ζητάει ανθρωπιστική βοήθεια αν παραμένει σιωπηλή όταν υπάρχουν ε, βόμβες ε, από τον ουρανό. Οι συνάδελφοι θέλουν να τα σπάσουν με τη Χαμάς. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στη Γάζα, θα δείτε την κατάσταση και θα δείτε γιατί κερδίζει η Χαμάς. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να βοηθήσει κανείς ε, το Ισραήλ ή τους Παλαιστινίους. Και ε, η άμεση κατάβαση του πυρός είναι μόνο ένα απόλυτο απαραίτητο βήμα. Ο κύριος Μπέρκ. Είναι σαφές ότι τα μέρη που συμμετέχουν στη σύραξη δεν συμμορφώνουν το διεθνές δίκαιο. Και ο άμαχος πληθυσμός της Γάζας πληρώνει το βαρύ τίμημα. Πρέπει να είναι κανείς υπόλογος στο διεθνές δίκαιο. Δεν γίνεται σεβαστά αρχές του πολέμου για αναλογικότητα και μη δικαιωματική χειρίση. Θα πρέπει λοιπόν η αναλογικότητα να επικρατήσει. Η ισχύ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι ανάλογη της βίας την οποία να ανταποκρίνεται. Η Χαμάς ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ναι. Αλλά η Ισραηλινή αντίδραση ήταν δυσανάλογη, κατά την άποψή μου. Δείτε τους αριθμούς. Πάνω από 900 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν. Πολύ λιγότεροι Ισραηλινοί. Το Ισραήλ θα πρέπει να απομειστεί τις ευθύνες του και θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ανάλογη δύναμη και συμμορφώνει το διεθνέ δίκαιο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε βέβαια ότι η Χαμά εξακολουθεί να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να, να μην απαρνιέται την ένοπλο, τον ένοπλο αγώνα, αλλά ε, με συνέπεια η Χαμά δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξη του Ισραήλ. Η Χαμά και άλλε παλαιστινιακέ ένοπλε δυνάμει θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο λαό του Νοτιού Ισραήλ έχει δικαίωμα να ζει άνευ βομβαρδισμών. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Μλάντενοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι όσοι παρατηρούν τη σύραξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπαίνουν στον πειρασμό να σηκώσουν τα χέρια στον αέρα και να ουρλιάξουν με απελπισία. Δεν πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό. Δοκιμάστε τον ανθρωπισμό μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής λύσης άνευ των βομβαρδισμών από πλευρά Ισραήλ. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχει διαρκή λύση χωρί να υπάρξει διέλευση ανθρωπιστική βοήθεια προ την Γάζα. Και ο πρόεδρο Πέρε σωστά το είπε. Η Γάζα θα πρέπει να ανοιχτεί για βοήθεια και δεν θα πρέπει να είναι κλεισμένη για τι ρουκέτε. Αυτό είναι η πεμπτουσία του θέματο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε στο θα του πω άντε και μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Το Κοινοβούλιο καταρχά μπορεί να φέρει τι δύο πλευρέ να συνομιλήσουν. Πρέπει να υποστηρίξουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προσπάθειε που καταβάλουν. Τρίτον, να υποστηρίξουμε και την Αιγυπτιακή προσπάθεια για διαπραγματεύσει. Αυτή είναι η μόνη διέξοδο, πιστεύω, που θα οδηγήσει σε μια λύση και κατάπαυση του πυρό. Κάτι για το οποίο ελπίζουμε όλοι. Ευχαριστούμε. Για Το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι ε, ότι μόνο εμείς είμαστε εξοργισμένοι από τις εξελίξεις στη Γάζα αλλά η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και αυτή είναι αγανακτισμένη από τον ε, πόνο των πολιτών στη Γάζα και από τον διαρκή αποκλεισμό. Έχουμε την ε, τρομοκράτηση ε, των αθών, κυρίως ε, των παιδιών και των γυναικών από τους Ισραηλινούς. Η παγκόσμια κοινότητα ζητάει την άμεση κατάβαυση του πυρός, αλλά προσκρούει σε ότα μία κόντων. Και ας μην ξεχνάμε, το Ισραήλ σε τελική ανάλυση θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε το Ισραήλ θα χάσει οποιαδήποτε υποστήριξη χέρι ακόμα από τη διεθνή κοινότητα. Δυστυχώ, Δυστυχώς ε, το ψήφισμα των ΗΕ είναι μονομερές ε, και είναι λυπηρό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ακόμα το ρόλο της. Ίσως αν λάβει στεναρότερα μέτρα από αυτά που έλαβε μέχρι τώρα ε, να τα πάει καλύτερα. Δεν πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας. Έχουμε κύρος, είμαστε σημαντικός εμπορικός εταίρος και χρηματοδότης σε αυτήν την περιοχή, άρα δηλαδή είμαστε σε θέση να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο.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 Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι αποδεκτό και μπορεί κανεί να το αιτιολογήσει με βάση το διεθνέ δίκαιο ότι για να εξωτρώσει κανεί τη χαμάσα το κράτο του Ισραήλ, μπορεί ε, δικαιούται να ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία τρομοκρατία και παραβίαση των συνθήκων των Ηνωμένων Εθνών ε, απέναντι όλα αυτά σε εγκλωβισμένου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπου. Και αυτά μπορούν να γίνονται ε, αγνοώντα τι δικέ μα αρχέ τη δημοκρατία. Το λόμπι των Ισραηλινών είναι τόσο τόσο ισχυρό έτσι ώστε ε, να καλεί την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να παραμένουν αδρανείς, αδρανείς και απλά να παρακολουθούν τις φρικαλαιότητες. Εάν οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι, τότε όλοι μας θα πρέπει την ελληνική κυβέρνηση να την πενέσουμε να πούμε πολύ καλά κάνατε, θαραλέει που μπήκατε στη Γάζα. Αν όμως είναι όχι, τότε θα πρέπει να καταδικάσουμε κατά κάθετα και αποφασιστικά το Ισραήλ να λάβουμε ταχύτατα αποφασιστικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών κυρώσεων έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή στη Γάζα και τώρα και για το μέλλον. Και ε, διαφωνώ κάθετα με τον Υπουργό Εξωτερικών που έφυγε, που είπε προηγουμένω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Κύρκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξελέγει εδώ και 25 χρόνια στο Κοινοβούλιο και είναι η σημαντικότερη συζήτηση στην οποία έχω συμμετάσχει. Κυρία Επίτροπε, ελπίζω να ακούσατε προσεκτικότατα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το βράδυ και το Κοινοβούλιο σήμερα. Ελπίζω να απαντήσετε στη συζήτησή σα και να πείτε ότι αντίθετα από τον Υπουργό Σβάτσεμπεργκ, ότι η ηθική πίεση μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον επιτιθέμενο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ισραηλινό λαό είναι ένα τίμιο λαό που έχει υποφέρει τα πάνδυνα επί αιώνε σε αυτή την Ήπειρο. Θα καταλάβει ο λαό τη σύστασή σα στο Συμβούλιο Υπουργών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσύρει αδίποτε επαφή, σταματά δίποτε επαφή με τις ελληνικές αρχές μέχρι ότου σταματήσουν τους βομβαρδισμούς. Ευχαριστούμε κύριε Μπίσλη. Το λόγο. Έχει ο ναι. κύριος Μασίπ για ένα λεπτό θα πρέπει να πούμε ομόφωνα στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να μας αφήσει να δράσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε τρόφιμα στο λαό αυτό και να τονίσουμε ότι η συμπεριφορά τους θα έχει επίπτωση σχέση με την Ευρώπη. Επίσης, Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αξίες μας, τις αξίες αλληλεγγύης της Ευρώπης, που θα πρέπει να είναι αποφασιστική σε αυτή την σύραξη. Τίποτα παραπάνω και σας ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι στο ψήφισμά μας επανειλημμένα αναφέρεται και υπογραμμίζεται μάλιστα ότι έχουμε αναβάλει, έχουμε παγώσει τη συμφωνία μας, τη διαδικασία για αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Ελπίζω λοιπόν να, να μην συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και business as usual. Δεύτερον, το Ισραήλ ποτέ, μα ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στι υποσχέσει που έδωσε. Δεν υπήρξε κατάπαυση του πυρό, διότι το Ισραήλ δεν ήρε τον αποκλεισμό του. Και το σημαντικό που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι μετά από αυτά που είχε υποσχεθεί το Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς, τι έγινε. Ο ρυθμός δημιουργίας επικισμών αυξήθηκε. Οπότε ποτέ δεν είχαν δημιουργηθεί τόσοι πολλοί επικισμοί κατά το παρελθόν. Σαν μανιτάρια φυτρώνουν εδώ και εκεί. Και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την Χαμάς να συμμορφωθεί με τους κανόνες μας αν δεν συμμορφωθεί και το Ισραήλ να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έδωσε. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Τώρα το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Στασνή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χθες Είχαμε κοινή αντιπροσωπεία, συνεδρίαση τη αντιπροσωπεία Παλαιστινίων και Ζαλινών. Φανταστείτε τώρα συνέστημα, ένταση, κατηγορίε και προτινόμενε λύσει μετά από 18 μέρε πολέμου στη Γάζα. Και περίπου χίλιου νεκρού. Γεγονό. Το Ισραήλ μετά από 8 χρόνια αναμονή αφού δέχτηκε περίπου 8.000 πυράβλους που τρομοκράτησαν περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους σύνορα με τη Γάζα, τελικά έχασε την υπομονή του Ισραήλ και άρχισε να προσπαθεί να πετύχει ασφάλεια για τους πολίτες. Δικαίωμά του είναι. Και υποχρέωση έχει το Ισραήλ για κάτι τέτοιο. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και είναι ο καθαρός ένοχος. Και είναι και βάρος για τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα. Η λύση είναι στα χέρια αναζωογονημένου κουαρτέτου. Και πρέπει να διπλασιαστούν οι προσπάθειες μεταξύ της νέας κυβερνήσεως των ΗΠΑ και της πλέον ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω προτεραιότητα της Προεδρίας και την άμεσο ενεργό προσπάθεια που κατέβαλαν στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Στάζνη. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σύραξη αυτή που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια βασίζεται σε εδαφικά προβλήματα αλλά και σε πολιτιστικά. Η λύση θα ήταν ένα Ισραηλινό κράτος δίπλα από ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό. Αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένοπλες επιθέσεις για να υπάρξει ένα βιωτικό επίπεδο αξιοπρεπές πρέπει να έχουν οι Παλαιστίνοι να αρνηθούν τον ένοπλο αγώνα και να ασχολούνται μάλλον με τη δημιουργία ενός κανονικού πολιτικού περιβάλλοντος προωθώντας πολιτικούς που προτιμούν τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Ντεμπρούν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ καταδικάζω την Ισραηλινή επίθεση στην Γάζα και εκφράζω και εγώ την αλληλεγγύη μου με τον λαό της. Είναι κρίμα που ακούσαμε ότι τα ΟΗΕ μπορεί να κάνει, λίγα μπορεί να κάνει, αλλά θα, το, ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα είναι να παγώσουμε κάθε σχέση με το Ισραήλ μέχρι να συμμορφωθεί με, το, με τη διεθνή νομοθεσία. Η συλλογική αυτή τιμωρία που επιβάλλει το Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας και που γίνεται με επίθεση ενός σύγχρονου στρατού σε έναν λαό που ήδη έχει υποφέρει πολλά από, την, από τον αποκλεισμό του είναι κάτι το τρομερό. Πρέπει να είναι σαφές ότι τα κύρια θύματα είναι ο αθώος λαός της Γάζας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεκέρτη. Ευχαριστώ. Με ανησυχία παρατηρούμε τα τεκτενόμενα στη Γάζα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Χαμάς προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Όμως καμιά από τις δύο πλευρές σε αυτή τη σύραξη δεν, έχουν δεν έχει υπόψη την ειρήνη. Η κάθε πλευρά έχει υπόψη τα δικά της συμφέροντα. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να συμφωνήσει να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος και το Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβουν. Πρέπει να τερματιστεί αυτό ο πόλεμο. Ο στρατό θα πρέπει να επιστρέψει στα στρατόπεδα και θα πρέπει η Χαμά να πάψει να εκτοξεύει πυράβλου κατά του Ισραήλ. Επίση πρέπει να προσφέρουμε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στου αμάχου ε, και στου τραυματισμένου. Προφανώ 3.000 ε, άμαχοι έχουν τραυματιστεί. Πρέπει η χώρα να επιστρέψει στην καθημερινή ομαλή ζωή και υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα που είναι σημαντικό. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριο Τιούρι, παρακαλώ. Yes, Mr. Ναι κύριε Σβόβοντα, παρακαλώ εσείς. Πρόεδρε, να σας ρωτήσω το εξή Έχουμε ακόμα και τη συζήτηση για το φυσικό αέριο σήμερα και περιμένουμε εμεί εδώ. Δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, αλλά και η συζήτηση για το φυσικό αέριο που είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Έχει αποσυρθεί, έχει διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη. Τι γίνεται. Το έχω υπόψη μου, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει. Λοιπόν, για ένα λεπτό, ο κύριος Γιώργη, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών της Προεδρίας ήταν πολύ απογοητευτική για μένα. Όλες οι ελπίδες μας βρίσκονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό γιατί, διότι ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς. Αν αναμείνουμε και ακόμα μια εβδομάδα θα φτάσουμε στους 1500 νεκρούς. Είναι δύσκολο να συζητήσει κανείς με τη Χαμάς. Είναι οργάνωση που έχει εγγραφεί στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Όμως το Ισραήλ είναι φίλος μας, εταίρος μας, σημαντικό μέλος της διεθνούς κοινότητας και πρέπει να παραμείνει και να σέβεται τους διεθνείς κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αν αποτύχει να το κάνει αυτό, τότε οι φίλοι και εταίροι του Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση να καταδικάσουν αυτέ τι πράξει του Ισραήλ και να υιοθετήσουν και κυρώσει. Πρόεδρο, καταλήγουμε τώρα σε αυτό τον ε, κύκλο και έχουμε τώρα την Επίτροπο που θα παρέμβει. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη γιατί ήταν πολύ μακρά η συζήτηση. Καταρχήν, να σα πω ότι ω μέλο ε, του κουαρτέτου της Μέσης Ανατολής εδώ και τέσσερα χρόνια μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να παίξει αλλά φυσικά δεν έχει τον ισχυρότερο ρόλο. Και αυτό φυσικά μας δημιουργεί απόγνωση, ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες στιγμές, όπου θα θέλαμε να πετύχουμε αμέσω μια βιώσιμη και διαρκή κατάπαυση του πυρός όπως προτείναμε, αλλά όπου δυστυχώς δεν μπορεί να επιτευχθεί τόσο γρήγορα. Αν Θα ήθελα να σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πηγές της Αιγύπτου που πρόσχεται στις διαβροματευτικές αποστολές δείχνουν ότι ε, η ΑΜΑΣ αντιδρά θετικά στην τελευταία Αιγυπτιακή πρόταση. Δεν ξέρω αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου της ΑΜΑΣ το απόγευμα στις 8. Φαίνεται πως κάπως προχωράνε τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει αυτό επιθυμούμε όλοι και ευχόμαστε. Να σας πω επίσης ότι με όλη την απόγνωση δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από ότι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ειρήνη. Και αυτό κάνουμε. Εγώ είμαι αφοσιωμένη σε αυτό. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο από κοινού και επίσης πρέπει να βοηθήσουμε τις προσπάθειες ε, της Παλαιστινιακής εμφυλίωσης γιατί μόνο τότε θα είναι δυνατόν να αποφύγουμε αυτή την ανομαλία της Γάζας. Βεβαίω, φυσικά, από τη στιγμή που υπάρχει η κατάπαυση πυρό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε τι βασικέ υπηρεσίε στον πληθυσμό, που τόσο άσχημα έχουν διακοπεί. Αυτό όμω που είναι πρωταρχικό αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει οι καταστροφές και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στην ανακοδόμηση και στη βιώσιμη ειρήνη.